was in a good mood. Um, well, that I wouldn't say. Buenos días. Monsieur. Muy buenos días. Good morning, everybody. Calmeda. Ε, ελπίζω οι διακοπές του Πάσχα να ήταν ευχάριστες και θετικές για όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής μας και να είμαστε κατά συνέπεια έτοιμοι για να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Όπως πάντα έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ημερήσια διάταξη. Θα σας παρακαλούσα εξ αρχής να συνεργαστούμε ούτε, ούτως ώστε να την προχωρήσουμε και αποτελεσματικά και γρήγορα. Το πρώτο θέμα που έχουμε μπροστά μας είναι η έγκριση της μερίσιας διάταξης. Να σας ε, αναφέρω ότι το σημείο 8 η έκθεση της κυρίας Γκάλ δηλαδή για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα αναβληθεί. Διότι η συγγήτρια δεν είναι παρούσα σε αυτή τη συνάντησή μας. Το ίδιο και το σημείο 19 για την οδηγία για την έκθεση Μωράες για τους δικαιού, την επέκταση του πεδίου εφαρμογή οδηγίας 109 του 2003 για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Εάν δεν έχετε κάποια άλλη παρατήρηση, εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Εγώ δεν έχω να σας κάνω ανακοινώσει. Πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Μου αναφέρουν ότι αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις Για τα πρακτικά μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ότι εγκρίθηκαν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Προχωρούμε στο σημείο 4 που αφορά στη δημιουργία ενός ε, γραφείου αξιωματικών συνδέσμων σε θέματα μετανάστευσης. Ο στόχος είναι η παρουσίαση της τροποποιημένης πρότασης. Ο κ. Δίας Δεμέρα είναι ο εισηγητής. Έχουμε μαζί μας τον κ. Μπράντλεϊ, εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας, Πριν ακούσουμε τον εισηγητή, ίσως θα ήταν σκόπιμο να ακούσουμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας. Τον κύριο Μπράντλι Είναι εδώ. Θέλει το λόγο. Θέλετε το λόγο κύριε Μπράντλι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην επιστολή σας στις 5 Μαρτίου ζητήσατε, θέστε μία ερώτηση που δεν είναι απλή. Θα σας πω γιατί. Και η συνθήκη αλλά και η νομολογία δεν δίνουν σαφείς οδηγίες για αυτό που ρωτάτε. Εσείς μιλάτε για, τον, για τη χρήση του όρου παράνομη μετανάστευση στη συνθήκη ή αντί για την ε, λάθρο μετανάστευση ή μη τακτοποιημένη μετανάστευση άλλους λόγους που έχουν λιγότερο βάρος. Το πρόβλημα είναι το εξή. Πρώτον, η μη τακτοποιημενη μεταναστευση αλλους λογους που εχουν λιγοτερο βαρος το προβλημα ειναι το εξης πρωτον η ορολογια της συνθήκης δεν τροποποιήθηκε με τη συνθήκη της Λισαμβόνας σε κάποιες γλώσσες τουλάχιστον. Σε ορισμένες χρησιμοποιείται η νέα ορολογία. Σε ορισμένες διατυπώσεις χρησιμοποιείται η παλιά. Επίσης, και μετά τις ορολογίες, μετά τι ε, αλλαγέ δεν έχει ενοποιηθεί η ορολογία σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές. Ξεκινούμε με την αγγλική εκδοχή. Ο όρος illegal immigration χρησιμοποιείται σε δύο διατάξεις. Στο 179 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης που είναι η νομική βάση του σχεδίου κανονισμού του οποίου είναι εισηγητής ο κ. Δίας Ντενέρα. Το 79.1 χρησιμοποιεί τον όρο αυτό για να δίνει μια γενική περιγραφή στους σκοπούς μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και την πρόληψη και την ενίσχυση συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και δια, ε, ατόμων. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται στο 79.2 που αναφέρει τα ειδικά μέτρα που μπορεί να υιοθετήσει ο νομοθέτης στον τομέα αυτό. Η παράγραφος Γ μίλα για μέτρα που αφορούν την παράνομη μετανάστευση, illegal immigration και την μη εγκεκριμένη παραμονή. Με άλλα λόγια, ο όρος παράνομη μετανάστευση στην πρώτη διάταξη του 79.1 έχει γενικό περιεχόμενο για κάθε μορφή μετανάστευσης που δεν τηρεί τις εφαρμοστές διατάξεις. Αυτό καλύπτει τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, οι οποίες πολίτες τρίτων χωρών μπορεί να βρεθούν μη τακτοποιημένοι στο εσωτερικό της Ένωσης και καλύπτει όσους εισέρχονται παράνομα με πλαστά έγγραφα, όσους έρχονται, εισέρχονται νόμιμα, αλλά ξεπερνούν το όριο παραμονής τους και όσους δεν λαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα. Ο όρος λοιπόν, illegality, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές. Στα ισπανικά είναι η illegal, στα γαλλικά legal, το ίδιο πράγμα σε όλες τις γλώσσες. Αυτό δεν ισχύει, <clears throat> ωστόσο, σε ό,τι αφορά το 79-2Γ. Η διάταξη αυτή σε όλες τις εκδοχές που είδαμε διακρίνει μεταξύ δύο διαφορετικών μορφών παράνομης παρουσίας, μη, μη νόμιμης παρουσίας. Το ένα στα αγγλικά είναι illegal immigration και unauthorized residence, αλλά δεν χρησιμοποιείται ο όρος illegal στην, στο ουσιαστικό ε, immigration. Αλλού χρησιμοποιείται ο όρος clandestine για την είσοδο και unauthorized για την παραμονή. Σε άλλες εκδοχές ισχύει το ανάποδο. Κατά την άποψή μας, Πρόεδρε, όταν υιοθετούνται συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης και παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, μπορούμε να χρησιμοποιούμε διαφορετική ορολογία από αυτή που χρησιμοποιεί το 79.2 γάμα, εφόσον γλωσσικά στέκει και ο όρος που χρησιμοποιείται το περιεχόμενο του όρου που χρησιμοποιείται ορίζεται σωστά. Δηλαδή ο νομοθέτης θα μπορούσε να μην χρησιμοποιεί τον όρο παράνομη, illegal μετανάστευση για την α ή β παράτυπη παρουσία πολιτών τρίτων χωρών στο ιστορικό της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, όταν το μέτρο που για το οποίο αναφορούμε χρησιμοποιεί τον όρο παράνομη μετανάστευση, illegal ε, immigration, με τον ευρύτερο όρο του 79.1, καλό θα ήταν κατά την απόψή μας να τηρήσουμε την διατύπωση αυτή. Γιατί αυτό που μετράει κυρίως είναι ε, η ασφάλεια δικαίου και όχι τόσο η συνέπεια στην οδολογία. Επιπλέον, το 79.1 όπως σας είπα χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο illegal για, σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές Τώρα για την τροποποίηση του κανονισμού 377 του 2004 ε, χρησιμοποιείται ο όρος illegal immigration, παράνομη μετανάστευση, μία φορά. Όταν μιλά για την έκδοχη του άρθρου 6 για την αναφορά θεμάτων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση. Το άρθρο 1.1 του κανονισμού διακρίνει άλλωστε μεταξύ της παράνομης μετανάστευσης και τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Αν χρησιμοποιούμε διαφορετικό όρο για το illegal immigration στην διάταξη αυτή, δημιουργεί σύγχυση. Γιατί δεν ξέρεις τι θα κάνεις με τον όρο μη εγκεκριμένη παραμονή. Αυτό που αναφέρει το 79 2 γάμα δηλαδή. Συνοψίζοντας, στον κανονισμό 377 ο όρος καλύπτει κάθε μορφή παράνομης μετανάστευσης και κατά την άποψή μας δεν θα ήταν σωστό να χρησιμοποιηθεί ο όρος αυτός παράνομη τώρα. Αντίθετα, θα έπρεπε να μπορούμε να διαφοροποιηθούμε στις άλλες περισσότερο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν σας διαφώτισα, είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Bradley. Vamos a escuchar ahora. Muy Θα ακούσουμε τον κύριο Δίας Μέρα και μετά θα γίνει ένας γύρος παρεμβάσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Μπράντλη και την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου που απάντησαν στο ερώτημά σας. Τους ευχαριστώ δε και για την προσπάθεια που κατέβαλαν να ερμηνεύσουν νομικά τον κανονισμό για το θέμα που θέσαμε. Το αν ήταν νομικά ορθό να χρησιμοποιούμε τον όρο, τον όρο illegal ή κάποιον άλλο όρο. <coughs> Είναι γεγονό ότι έχουμε μπροστά μας κάτι που ξεπερνά τη νομική διάσταση του θέματος. Πρόκειται για μία κατάσταση, γενικευμένη άποψη που έχει να κάνει το εξή. Η νέα φωνή του Κοινοβουλίου μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι μία πολύ πιο δυνατή φωνή, μία φωνή που πρέπει να ακούγεται Για παράδειγμα, τη δύναμη της φωνή αυτής θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με την τροποποίηση αυτή του, συμφώνησε με την τροποποίηση του κανονισμού αυτού σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα συμφώνησαν στο Συμβούλιο, γιατί προφανώ ήταν ένα θέμα ίσονο σημασία, χωρίς πολλά προβλήματα. Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, και η Επιτροπή έχει τέσσερις συνεδριάσεις έντονης δουλειάς και μία συνάντηση του εισηγητή με τους σκιώδεις για το ίδιο θέμα. Κατά την άποψή μας λοιπόν, δεν είναι ίσονος σημασίας το αν θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο παράνομο ή μη νόμιμο, κατά την άποψη δική μας και κατά την άποψη και της Επιτροπής γιατί και η Επιτροπή μας υποστηρίζει. Η Επιτροπή απεχθάνεται τη χρήση του όρου παράνομος, illegal, όταν αναφέρεται σε άτομα που κατά την άποψή μας είναι χωρίς νόμιμα έγγραφα. Πάντω, λέει ο κύριος Μπραντρί ότι το άρθρο 79.1 τη συνθήκη Λειτουργία Ένωση χρησιμοποιείται για την κάλυψη όλων εκείνων των μορφών μετανάστευση που για τον α ή β λόγο δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστές διατάξεις του νόμου. Αυτή είναι η ισχύουσα, η κυρίαρχη ερμηνεία των νομικών υπηρεσιών για το 79.1. Επίσης όμως ο κύριος Μπλάτλεϊ μας είπε ότι το 79.2 το άρθρο 2 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης ε, ο όρος εκεί ε, αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στις συνέπειες της παράνομης εισαγωγικά εισόδου που είναι ωστόσο κάτι διακεκριμένο, κάτι ξεχωριστό από την μη εγκεκριμένη παραμονή. Περίπλοκο είναι, αλλά αυτό που, ήθελε να, που θέλει να πει η έκθεση του Κοινοβουλίου είναι ότι εν γέννη πρέπει να τηρούμε το 79.1 και μόνο σε πολύ επιμέρους συγκεκριμένα θέματα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η διάκριση του παράτνομους ε, που μας επιτρέπει το 79.2. Αυτή η μακρά παρέμβαση που κάνω, πού μας οδηγεί στο εξής. Εγώ θα μιλήσω εκ νέου με τους σκιώδεις εισηγητές, ούτως ώστε λαμβάνοντας υπόψη, όπως πάντα σχεδόν κάνουμε, την ε, άποψη της νομικής υπηρεσίας του σώματος, θα μπορέσουμε να βρούμε μία ενδεδειγμένη διατύπωση που κατά πάση πιθανότητα θα είναι η χρήση και των δύο όρων. Δηλαδή και illegal και irregular ή και illegal και clandestine. Αφού δούμε τι αναφέρει το 79.1, τι αναφέρει το 79.2 στις διάφορες εκδοχές και να σας δώσω και ένα παράδειγμα πολύ επίκαιρο. Η πιο πρόσφατη νομοθεσία και πιο σύγχρονη νομοθεσία για την μετανάστευση είναι η Ισπανική μεταξύ των 27 του Νοεμβρίου. Όπως ξέρετε, ο νόμος αυτός τι έκφραση χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί τον όρο παράτυπη ή τον όρο παράνημη. Η απάντηση είναι εκπληκτική. Σας εκπλήσει. Όπως ακριβώ το 79 και 2. Χρησιμοποιούνται και οι δύο εκφράσεις στο νόμο. Και ο όρος irregular, irregular και illegal. Λίγο πιο συχνά χρησιμοποιείται ο όρος παράτυπος και όχι παράνομος. Άρα το θέμα είναι ένα θέμα που δεν έχει λυθεί και που θα πρέπει για να το λύσουμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ φαντασία. Πρέπει να είναι σαφές ωστόσο ότι η θέση μας είναι περισσότερο στην χρήση του όρου irregular παρά στη χρήση του όρου illegal. Πέραν αυτού, πρόεδρε, έχουν υποβληθεί 24 τροπολογίες είχαμε συζητήσει τις τοπολογίες και σας έδωσα ένα φύλλο, αυτό που, που περιλαμβάνει τις τοπολογίες που μπορώ να δεχτώ και τις τοπολογίες που δεν μπορώ να δεχτώ. Ανεξάρτητα λοιπόν το ότι η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι εγώ είμαι ανοιχτό σε νέες ε, συμφωνίες, θα μπορούσαμε, και αυτή είναι η πρόταση που κάνω και προς την Επιτροπή Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε να γίνει μια προσπάθεια ψηφοφορίας στις 27-28 Απριλίου στις συνεδρίες της Επιτροπής. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Πριν τους συναδέλφους να ακούσουμε σύντομα την άποψη του Εδρές και της Επιτροπής. Ο κύριος Ντόμπο από την Επιτροπή. Θέλει το λόγο. Η κυρία. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τέλο πάντων. Εσείς. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία για την παρέμβασή της. Και όσον αφορά την νομική ασφάλεια, όλοι σκεφτόμαστε πως είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται η γενικότερο όρο της παράνομης μετανάστευσης, illegal immigration, ώστε να αποφευχθούν ε, οι παρεξηγήσεις. Σας ευχαριστώ. Κύριε ευχαριστώ στο Συμβούλιο εξετάσαμε την πρόταση της Επιτροπής και την είδαμε με θετικό πνεύμα, με κάποιες μικρές τροποποίησεις, χωρίς ουσιαστικά του ουσιαστικό τόσο. Κατά την άποψή μας η πρόταση αυτή βελτιώνει την πρακτική συνεργασία των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, ένας ε, επιθυμητός στόχος με την γενική αυτή υποστήριξη λοιπόν προς την πρόταση επιστοπής θα ήθελα να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό με το Κοινοβούλιο τις συζητήσεις για τις τροπολογίες στον κανονισμό. Να πω προς την να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία της Επιτροπής για την έκθεσή της. Θα τη μεταφέρουμε στο Συμβούλιο. Εκ πρώτης όψεως ωστόσο μου φαίνεται θεμελιωμένη και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ, ήσασταν σύντομοι. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μας έδωσε γνωμοδότηση η νομική υπηρεσία, αλλά η γνωμοδότηση αυτή από τη νομική υπηρεσία αφορά το θέμα της νομολογίας του τι είναι νόμιμο. Εμείς όμως είμαστε και πολιτικοί που πρέπει να λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις. Τι σημαίνει παράνομος, illegal, σε πολιτικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πέρα από το σωστό όρο στο δίκαιο. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ ανθρώπων που εισέρχονται παράνομα, υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών που εισέρχονται παράνομα και αυτών που εισέρχονται νόμιμα. Αλλά ε, παραμένουν και πέραν της νόμιμης εξουσιοδότησης. Ε, επίσης, ε, πολλές φορές θα πρέπει να δούμε τι συνιστά αξιόπινη πράξη. Ε, Ε, αξιόπινη πράξη δεν είναι η παράνομη παρανομή, η παράνομη είσοδος σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν συνιστά παντού αξιόπινη πράξη. Ε, σε ορισμένα ναι, αλλά όχι σε όλα. Οπότε δεν πρόκειται για πραγματική παρανομία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε αυτή την πολιτική απόφαση, να πάρουμε μια απόφαση που θα εκφράζει τις πολιτικές μας απόψεις και γι' αυτό η ομάδα μου προτιμά την διατύπωση ε, irregular και όχι illegal. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριος Μπρόγκς. Αυτό που λέμε ότι μπορεί η παρανομία να είναι παράταση πέραν της νόμης παραμονής, η παράνομη είσοδος ή παραμονή μετά την απόρριψη του εξέτησης ασύλου. Δηλαδή είναι κάποιος παρόν, διαμένει παράνομα σε μια χώρα ε, η ληστεία ας πούμε. Μπορεί να γίνει επειδή παίρνω κάτι χωρίς άδεια ή επειδή μου δάνεισαν κάτι και, αλλά εγώ δεν το επέστρεψα ποτέ ή παίρνω κάτι και παράλληλα το ζητάω και όταν απορρίπτεται το αίτημα εξακολουθώ να κρατώ το αντικείμενο, το προϊόν. Πρόκειται για κλοπή. Ε, δεν λέω ότι είναι ίδια η κατηγορία, αλλά υπάρχει μια αναλογία. Θα πρέπει να δούμε το, τη γλωσσική διατύπωση. Αυτό είναι μια ιδέα που ο George Orwell θα περιέγραφε ως έλεγχο της σκέψης. Όταν ελέγχονται οι γλώσσες που μιλούν οι άνθρωποι, ελέγχονται και οι σκέψεις τους. Αυτοί που θέλουν να σκέφτονται ελεύθερα στην Επιτροπή πρέπει να επιλέξουν τη δική τους διατύπωση όπως θεωρούν ε, αρμόζουσα στη δική τους γλώσσα. Ευχαριστώ. Κύριος Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ζητήσω ε, ένα αντίγραφο της νομοδότησης νομικής υπηρεσίας. Αν υπάρχει ε, έγγραφο, θα ήθελα πολύ να διαβάσω αυτή την επιχειρηματολογία. Τώρα, μετά από αυτά που ακούσαμε από την νομική υπηρεσία, νομίζω ότι υπάρχει εδώ σε ε, διπλό επίπεδο η συζήτηση σε νομικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Μετά από αυτά που μας είπε ο κύριος Μπράντλι, από νομικής άποψης δεν υπάρχει αμφιβολία και πρέπει να μιλούμε για illegal ε, ε, μετανάστευση. Από πολιτικής άποψης πολλές φορές ε, θέτουμε το ερώτημα αν είναι πολιτικά σωστό να μιλάμε για illegal ή αν θα πρέπει να επιλέξουμε την υπιότερη διατύπωση irregular. Αυτό είναι μια πολιτική αντιπαράθεση και κυρία Δίας πρέπει να διαφοροποιήσουμε σαφώς μεταξύ πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης. Σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να αποφασίσουμε ότι είναι λάθος πολιτικά να μιλήσουμε για illegal μετανάστευση. Αυτό που μας λέει σήμερα η νομική υπηρεσία είναι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας και η συνθήκη μας πολιτικά είναι λάθος. Εντάξει, θα πρέπει όμως να ε, ε, δούμε ότι τα νομικά μας κείμενα μιλούν για illegal, δεν μπορούμε να τα τροποποιήσουμε, άρα πρέπει να διατηρήσουμε τη διατύπωση illegal. Γιατί ακόμα και αν θεωρούμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να έχει ε, τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, όμως Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τις διατάξεις της συνθήκης. Και όταν πρόκειται για νομοθεσία, αλλάζοντας την έννοια illegal που υπάρχει στη συνθήκη, ούτως ώστε να γίνει politically correct, τότε στο τέλος θα δημιουργήσουμε σύγχυση, όπως άλλωστε σαφώς μας ετώνησε η νομική υπηρεσία. Ε, ε, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη λοιπόν, απευθύνω έκκληση στον εισηγητή να διατηρήσει τη νομική έννοια illegal επειδή δεν είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τις διατάξεις της συνθήκης. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διατύπωση. Η επίμετρον η Κομισιόν επίσης ε, μάλλον θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη λέξη illegal ως γενικότερη κατηγορία ενώ το Συμβούλιο επίσης συμφωνεί. Άρα δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί εμείς να διαφοροποιηθούμε. Ευχαριστώ. Madame Guillaume. Euh, να σύντομα, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Δίας Δεμέρα για τον διάλογο που ξεκίνησε με τους Σκιώδης, εκ των οποίων είμαι και εγώ μέρος. Και διαπίστωσα κατά τη διάρκεια αυτών των παρεμβάσεων πως το Κοινοβούλιο επ' αυτού του θέματος θα πρέπει να υπερασπιστεί μια ισχυρή θέση. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν από την νομική υπηρεσία και έπειτα από τους διάφορους συναδέλφους, Βλέπουμε σαφώς πως η συνέχιση της συζήτησης για το θέμα της ορολογίας θα είναι σκόπεμη και ευχαριστώ επίσης τον κύριο Τιάς Δεμέρα που πρότεινε κάτι τέτοιο, διότι ανάμεσα στους διάφορους νομικούς ορισμούς θα έχουμε να κάνουμε και μια πολιτική αξιολόγηση. Και πιστεύω και εγώ πως θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση Κατά την άποψή μου θα έλεγα ότι οι ορισμοί δεν είναι ουδέτεροι και προσωπικά είναι, όπως είπε και η κυρία Κέλλερ, να θεωρώ πιο σκόπιμη τη χρήση του όρου irregular ε, που μου φαίνεται πιο καλά, ε, πιο κατάλληλη μάλλον δεδομένων των ε, συνθήκων. Τώρα δεν ξέρω σε ποια στιγμή θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση αν και εσείς το κρίνετε απαραίτητο αλλά είμαι μεταξύ αυτών που έχουν καταθέσει τροπολογίες εκτός και πέρα από την ίδια την τροποποιημένη πρόταση που θα μπορούσαν να έρθουν σε ε, σύγκρουση με διάφορες άλλες λειτουργίες πιο άτυπες και θα ήθελα να δούμε μαζί πώς θα μπορέσουμε να εγκαταλείψουμε τις τροπολογίες που δεν χρειάζονται και να τηρήσουμε την νομική βάση που μας έχει προταθεί. Και τελευταία παρατήρηση σε σχέση με όλα αυτά. Κατανόησα ότι αυτή η τροποποιημένη πρόταση είναι η μόνη επί της οποίας μπορούμε να εκφραστούμε. Αλλά ακριβώς επειδή θέλουμε να μιλήσουμε και να αξιοποιήσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου, Ίσως θα έπρεπε να διαρωτηθούμε για το μέλλον, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαβούλευση, πέρα από τα όσα προτείνονται ω τροποποίηση. Δεν ξέρω αν έγινα σαφή, πάντω γενικά μιλώ υπέρ τη ενίσχυση των εξουσιών του Κοινοβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι δύσκολα ε, ε, θα ξεμπλέξουμε από μια συζήτηση αντιπαράθεσης ενιών. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν την ουσία της μετανάστευσης. Ε, δεν, θα, ε, δεν με πειράζει ε, ο όρος παράνομη μετανάστευση, αλλά παράνομη ε, γενικότερα όσον αφορά σε ανθρώπους. αν δεν θα αναφερόμουν ποτέ σε ένα μετανάστη ως παράνομο, παράνομος ως άνθρωπος, δηλαδή υπάρχουν παράνομοι ή ε, μη ρυθμισμένοι ή regular τέλο πάντων τρόποι εισόδου. Όμως η Επιτροπή έχει συμφωνήσει εδώ και χρόνια να αποφεύγει την ε, χρήση της έννοιας illegal ε, ως ε, επίθετο σε ανθρώπους. Νομίζω ότι και στην έκθεση μπορούμε να συνεχίσουμε ε, να χρησιμοποιούμε τη λέξη irregular. Αν μιλήσουμε για illegal migration, εντάξει, μπορούμε για να καλύψουμε και τις ε, σχετικές ε, προτάσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει το επίθετο illegal να αναφέρεται σε πρόσωπα. Δεν θέλω να μπω σε σημειολογικές παρατηρήσεις. Η ουσία νομίζω ότι είναι σημαντικότερη. Ευχαριστώ. Thank you. Creo que Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τον εισηγητή να ολοκληρώσει και να κάνει μια πρόταση για τα επόμενα βήματα σε σχέση με την πρότασή του. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ εκ νέου και το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και την κυρία Κίλε, τον κύριο Μπρόντσο, τον κύριο Μπουσούτιλ την κυρία Γιγιόμ, τη Σιλβή και τον κύριο Λαμπρινίδη για τις παρεμβάσεις τους που εμπλούτησαν την συζήτηση. Το πρώτο που ήθελα να επαναλάβω, Πρόεδρε, είναι ότι είμαι έτοιμος να συνεχίσω τις, το διάλογο και τις συζητήσεις. Και δεύτερον, να θέσω έναν χρονικό ορίζοντα για την διαπραγμάτευση αυτή. Αυτό θέλω να προτείνω. 27-28 Απριλίου για να αποτιμήσουμε σε πρώτη φάση πού είμαστε σύμφωνοι, πού διαφωνούμε για την έκθεση. Επίσης, πρέπει να κάνουμε κάτι και στο εσωτερικό των ομάδων μας. Για αυτό το σημειολογικό νομικό ζήτημα, που είναι και πολιτικό βεβαίως. Πρέπει να αποφασίσουμε στο περιθώριο των προσωπικών απόψεων, αξιοσέβαστες καθόλα, πρέπει ωστόσο να δεχθούμε και πολύ συχνά πιστεύω ότι έστω και αν διαφωνώ, πρέπει να ακούσω τις απόψεις της πολιτικής μου ομάδα. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πετύχω εγώ είναι να έχω μια πολιτική συζήτηση στη δική μου ομάδα για να δω κατά πόσον είναι προτιμότερη η σωστή και νομική έκφραση παράνομος ή η πολιτική έκφραση παράτυπος ή λάθρα, η regular clandestine. Αυτό είναι αναγκαίο πιστεύω, διότι είναι προφανώς ένα πολιτικό ζήτημα και αυτό πρέπει να συζητηθεί κατά την άποψή μου στο εσωτερικό των ομάδων. Και ό,τι αφορά τώρα την ουσία του θέματος, θέλω να πω κάτι μόνο. Ευχαριστώ την Σιλβή για τις τροπολογίες που έχει υποβάλει, θεμελιωμένες και εύλογες. Ο μόνος λόγος για την απόρριψη ορισμένων εξ αυτών είναι αυτό ακριβώς που μας είπε η ίδια, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που δεν μπορεί να τροποποιηθεί βάσει τις προτάσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Σε μελλοντικές εκθέσεις, ωστόσο, είναι δυνατό να υπησέλθουμε σε νέες διαστάσεις που είναι αντικείμενο κάποιων από των τροπολογιών της κυρίας Γκυγιόμ. Τελειώνοντας, Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή μας να λάβει θέση εν γέννη, όχι ξεκάθαρη, ως προς τις υπόλοιπες τροπολογίες. Είναι σημαντικό νομίζω να ακούσουμε τι λέει η Επιτροπή που γνωρίζει τις τροπολογίες μας. Θα ζητούσα λοιπόν από την Επιτροπή να λάβει θέση για τις τροπολογίες εκείνες που δεν έχουν να κάνουν με την πλούσια συζήτηση που είχαμε για τον όρο παράνομος, παράτυπος ε, Χωρί τι νόμιμε διατυπώσεις. Αυτά τα ολίγα, πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, λέει πρόεδρο. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να σημειώσουμε ότι η έκθεση της νομικής υπηρεσία που παρουσίασε ο κύριος Μπραντλή διανεμήθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Την έχετε λοιπόν στα χέρια σας κύριε Μπουσούτιλ. Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε την διατύπωση της Επιτροπής για τη, τους όρους που αναφέρονται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα για να απαντήσω στις ερωτήσεις του κ. Ντίας Δεμέρα. 28-29 θα γίνει η συζήτηση. Δέχομαι την πρότασή του να έχουμε μια πολιτική συζήτηση στις ε, πολιτικές ομάδες για το θέμα αυτό και με αυτά προχωρούμε στο, στο επόμενο σημείο στη μέση διάταξη, το σημείο 5. Συμφωνία μεταξύ Ένωσης Ισλανδίας και Νορβηγίας για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αποφάσεων του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση, την μάχη κατά της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Φόουλ από την Επιτροπή. You course. <laughs> What's spring? spring. So. So λοιπόν, την, η απόφαση του Συμβουλίου που είναι γνωστή και ως απόφαση πριν είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών εμείς θεωρούμε ότι μαζί με την παρουσίαση των βασικών στοιχείων της απόφασης και της κατάστασης για την εφαρμογή των αποφάσεων θα ήταν κάτι θετικό. Δίνω λοιπόν το λόγο Όχι, λέει η Διοκάπτειο μιλητής. Πριν δώσει το λόγο στον εισηγητή θα ακούσουμε την Επιτροπή. Πρώτα η Επιτροπή, μετά ο κύριος Μπουσούτιλ. Κύριε Φόουλ, έχετε το λόγο. Thank ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Αυτή η συμφωνία είναι σημαντική γιατί κατοπτρίζει το βάθος των σχέσεων μεταξύ ημών και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Εμείς στην Κομισιόν ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα δώσει την εγκρισή του για τη συμφωνία αυτή. Σύντομα, η στενή συνεργασία μεταξύ ημών και αυτών των δύο χωρών βασίζεται στην ε, Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που είναι το βασικό νομικό μέσο ε, που μας συνδέει. Αυτό σημαίνει βέβαια πως η Νορβηγία και η Ισλανδία έχουν εφαρμόσει την οδηγία για την προστασία των ε, δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων 9546 είναι μέλη του Σέγγεν και άρα είναι συνδεδεμένες και σέβονται τους κανόνες του Σέγγεν συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί αστυνομικής συνεργασίας, ενημέρωση Σέγγεν, το μελλοντικό σύστημα θεωρήσεων, το Frontex και άλλα συστήματα που συνδέονται με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, γιατί τα δικά του σύνορα είναι δικά μας εξωτερικά σύνορα και τούμπαλιν. Στο πλαίσιο αυτή της συνεργασίας με το σύστημα του Σέγγεν και οι δύο χώρες έχουν εφαρμόσει στον εθνικό τους νόμο, στην εθνική τους νομοθεσία, τις διατάξεις που αφορούν ε, την ε, αποκαλούμενη απόφαση πλαίσιο, τη ε, απόφαση πλαίσιο, καθώς και όλες τις διατάξεις που αφορούν τον τρίτο πυλώνα, όπως λεγόταν παλιότερα. Έχουν ειδικέ συμφωνίες με τη Eurojust, το Euro παλ και την ΣΕΠΑΡ ε, συνδεδεμένοι με το Ευρωπόλ έχουν ε, παρατηρητές εκεί και η Νορβηγία έχει και έναν εισαγγελέα που είναι τοποθετημένο στο Eurojust. Συμμετέχουν στον κανονισμό του Δουβλίνου καθώς και το σύστημα Eurodac που απορρέει από αυτό είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Σύμβαση του 1981 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το Πρωτόκολλο 2001, καθώς και τη σύσταση 8715 της Επιτροπής των Υπουργών για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας. Έχουν επίσης ε, τηρήσει τις απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων για την ε, δυνατότητα ανταλλαγής. Ε, ε, δεδομένων. Θέλουν να μπουν στο σύστημα πρόμα, να συμμετέχουν στο Σέγγεν χωρίς το πρόμα Είναι λιγότερο αποτελεσματικό για την καταπολέμηση των διασυνοριακών εγκλημάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω πως ε, μπορούν να αποτελέσουν τμήμα του συστήματος πρόμα και ελπίζω πως θα το κάνουν μια, δύο λόγια για, σε σχέση με το αίτημα του Προέδρου για το τι συμβαίνει στο σύστημα ΠΡΟΜ και πώς λειτουργεί. Οι αποφάσεις ΠΡΟΜ ρυθμίζουν ε, την ε, ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων διασυνοριακά όσον αφορά τις τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά και την αναζήτηση προφίλ DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και ούτω καθεξής. Τα κράτη-μέλη είχαν μέχρι τον Αύγουστο του 2009 για να εφαρμόσουν τι διατάξει που σχετίζονται με τέτοια γεγονότα για την πρόληψη τη τρομοκρατίας και έχουν μέχρι τι 26 του Αυγούστου του 2011 για να εφαρμόσουν τι διατάξει που αφορούν την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή στοιχείων. Τώρα, για να ξεκινήσει η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή στοιχείων θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προβούν στα εξή βήματα, δηλαδή να κοινοποιήσουν τον εθνικό του σύνδεσμο στο Συμβούλιο, να διευκρινίσουν του ε, φακέλου ανάλυση DNA προ το Συμβούλιο, να διευκρινίσουν διερευνήσουν επίσης τις ημερήσιες δυνατότητες ανάλυσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, να δουν να κοινοποιήσουν τα μέσα που χρησιμοποιούν και να εφαρμόσουν όλες τις απαιτήσεις ε, Προστασία δεδομένων πριν προβείουμε σε οποιαδήποτε ανταλλαγή στοιχείων. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αν πληρούνται όλε αυτέ οι προποθέσει. Και φυσικά θα πρέπει να ανταποκριθούν σε όλε τι τεχνικέ απαιτήσει όσον αφορά την αυτοποιημένη ανταλλαγή στοιχείων, συμπεριλαμβανομένη τη σύνθεση στην Εστέστα και στην εφαρμογή Ιουκάρης. Μην με ρωτήσετε παρακαλώ τι είναι αυτά όλα αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούνται σημαντικά για την, ανταλλαγή, την ασφαλή ανταλλαγή ε, στοιχείων. Τα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει, που έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτό το τομέα, βοηθούν τα υπόλοιπα με την προετοιμασία για την πληροφορική, γίνονται δοκιμαστικές ε, ε, δοκιμαστικά μάλλον λειτουργούν τα συστήματα, γίνονται επισκέψεις επιθεώρησης, γίνεται μια διαδικασία αξιολόγησης ε, στους ε, τομείς ε, του DNA και της καταγραφής των αυτοκινήτων, των πινακίδων των αυτοκινήτων και η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά την συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με τις απαιτήσεις για την ανταλλαγή των δεδομένων. Όλα αυτά τα συστήματα έχουν εγκριθεί για τα κρατημέλη όσον αφορά το DNA, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Σλοβενία σε σχέση με τα αποτυπώματα δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει. Ε, και σε σχέση με την καταγραφή των πινακίδων 7 από τους 27 Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, η Γαλλία και οι κατοχώρες τα εξή κράτη-μέλη θα υποστούν την αξιολόγηση στο δεύτερο ήμιση του 2020, DNA για το Βέλγιο, αποτυπώματα για την Βουλγαρία και την Γαλλία στο δεύτερο ήμιση του έτους και για τις πινακίδες αυτοκινήτων για τη Φιλανδία έγινε μια πρόσφατη εξολόγηση που ήταν επιτυχής. Και το δεύτερο ήμιση του έτους θα γίνει μια τέτοια εξολόγηση και για τη Σλοβενία Αυτή είναι η κατάσταση. Το σύστημα λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά και πιστεύουμε πως θα πρέπει να επεκταθεί στην Νορβηγία και την Ισλανδία είναι προς το συμφέρον του, αλλά είναι και προς το δικό μας συμφέρον να μην έχουμε αδύναμους κρίκους στην αλυσίδα του Σέγγεν και ελπίζουμε πως το σύστημα αυτό θα εγκριθεί και θα αρχίσει να ισχύει όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Thank you. Now we hear from the rapporteur. Ευχαριστώ. Και τώρα ο εισηγητή μα, ο κύριο Μπουσούτιλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φόλ για την πολύ λεπτομερή παρουσίαση που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε επί της ουσίας του φακέλου αυτού. Θα περιοριστώ σε τέσσερις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, θέλουμε να επεκτείνουμε την απόφαση Προύμ για να συμπεριλάβουμε την συμμετοχή Νορβηγίας και Ισλανδίας. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει προς εμάς η έκθεση. Εδώ η απάντηση που προτείνω στους συναδέλφους είναι να απαντήσουμε καταφατικά. Ναι, πρέπει να συμφωνήσουμε ε, στη συμμετοχή Ισλανδίας και Νορβηγίας στην απόφαση Προύμ. Δεύτερον, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από άποψη ουσίας, σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, προστασία δεδομένων, διαφοροποιούνται σε σχέση με τα ισχύοντα καθημάς. Ε, κατά τη γνώμη μου, θέλω όμως να μου επιβεβαιωθεί αυτό, υπάρχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως ισχύουν για μας. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά ε, σε σχέση με την Ισλανδία και την Νορβηγία. Τρίτον, είναι προς το στρατηγικό μας συμφέρον να πούμε ναι στην συμμετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στην απόφαση πριν. Εγώ θα έλεγα προς τους συναδέλφους ότι ναι, μας εξυπηρετεί. Γιατί αν συνεργαστούμε στην πάλι κατά της τρομοκρατίας δεν βοηθούμε μόνο τις ε, φίλες αυτές χώρες, ε, αλλά εξυπηρετούμε και τα ε, θέματα ασφαλείας των πολιτών μας. Τέλος, και εδώ θα ήθελα να μου επιβεβαιώσει η Κομισιόν, η Ισλανδία και η Νορβηγία από τεχνικής άποψης είναι έτοιμες. Υπάρχουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο κύριος Φόλ έδωσε κάποιες λεπτομέρειες ως προς αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιβεβαιώσει ότι πράγματι οι δύο χώρες είναι σε θέση να ε, προσχωρήσουν από τεχνικής άποψης. Αυτές είναι οι τέσσερις παρατηρήσεις μου κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ε, ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων αν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια από τους συναδέλφους, ποιος ζητεί το λόγο. εκπρόσωπος της Προεδρίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από πλευράς Προεδρίας του Συμβουλίου αυτό που καταρχάς θα θέλαμε είναι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φόλ για την πολύ λεπτομεριακή ανάλυση που έκανε. Δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε. Και απλά να επιβεβαιώσω αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μπουσούτιλ για την σπουδαιότητα της συμφωνίας αυτής. Το Συμβούλιο ομόφωνα έχει την άποψη ότι η συμφωνία αυτή είναι κάτι εξαιρετικά αναγκαίο που θα συμπληρώσει το πλαίσιο αυτό που γεωγραφικά δεν έχει πλέον όρια ε, μεταξύ Ισλανδίας και Σέγγεν. Ε, ε, ωστόσο παραμένει μία διάσταση αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας που με την ανταλλαγή αυτή των δεδομένων ενισχύεται σημαντικά εάν εφαρμοστεί η απόφαση αυτή και αν υπογραφεί η συμφωνία αυτή και εμπιτευτεί η ανταλλαγή δεδομένων θα είχαμε πετύχει κάτι πολύ χρήσιμο. Έθεσε μία ερώτηση ο κύριος Μπουσούτιλ για την τεχνική προπαρασκευή των δύο χωρών για την ένταξή τους στο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων. Εδώ υπάρχουν δύο συναφή μεταξύ τους θέματα. Πρώτον, το να προχωρήσει τεχνικά κάτι που δεν έχει την πολιτική επιβεβαίωση ακόμα, ούτε την νόμιμη έγκριση, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία, δημιουργεί κάποιους κινδύνους. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι εθνικές εξελίξεις, η κατάσταση στον τομέα της προστασίας ε, των δεδομένων και τα τεχνικά στοιχεία που μπορεί να διευκολύνουν την ανταλλαγή αυτή είναι πλήρης από πλευράς των χωρών αυτών, αλλά όπως όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία τεχνικής εξέτασης που θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μετά τη θέση ισχύ της συμφωνίας. Αυτά και ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Σχόλια. Όχι. Yes, please, Mr. Fall. Just the answer to... Να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ναι και στις δύο και συμφωνώ και απόλυτα με αυτό που είπε ο εκπρόσωπος Συμβουλίου. Υπάρχει μια, ένα πλήρες ε, σύστημα αξιολόγησης. όλο τόσο δείχνουν πως οι δύο χώρες είναι έτοιμες να αναλάβουν τις υποχρεώσει. Είναι παρόμοιες, είναι ίδιες με αυτές που έχουμε και θα ενισχυθεί σημαντικά το σύστημα του Σέγγεν εάν οι χώρες αυτές ενταχθούν στο σύστημα του ΠΡΙΜ. Ευχαριστώ. Αυτά προς το παρόν. Σημείο 6. Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ για την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΣΥΠΑ για σκοπούς της, ε, του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εδώ έχουμε στόχο να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τη νέα συμφωνία. οι συντονιστές ενημερώθηκαν στις 24 Μαρτίου από την Επιτροπή για το περιεχόμενο του νέου σχέδιου εντολής μακροχρόνιας συμφωνίας ε, Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την συμφωνία αυτή διαβίβασης δεδομένων χρηματοπιστικών ε, συναλλαγών. Το περιεχόμενο ωστόσο είναι ε, εμπιστευτικό και τα μέρη μπορούν να τα εξετάσουν μόνο υπό τη διαδικασία του εμπιστευτικού. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για την, ε, τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί με το νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Από ό,τι φαίνεται εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα ωστόσο θα ζητήσω από την εισηγήτριά μας την κυρία Χάνη Πλασάρτ να μας δώσει μια γενική εικόνα του θέματος. Ζανίν, έχετε το λόγο. Γενική... Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών προσπάθησα να βάλω κάποια τάξη σε όλα αυτά. Θα πρέπει να σας πω ότι αρχικά είχα μια θετική αντίδραση στην εντολή που μας παρουσίασε η Κομισιόν στις 24 Μαρτίου. Μετά κάπως ε, μπόρεσα να αναλύσω αυτές τις πληροφορίες και να σας, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν προσπαθεί να βρει καμιά εναλλακτική λύση. Δηλαδή πρέπει όντως από πρώτη όψης να δούμε πως αυτή η εντολή ανταποκρίνεται σε διάφορες απαιτήσεις του Κοινοβουλίου. Ωστόσο φοβούμε πως αυτό γίνεται σε πολύ επιφανειακό επίπεδο. Αυτή η εντολή λοιπόν αφορά την βράχη πρόθεσμη λύση των εφαρμοστικών θεμάτων αλλά όχι ε, την μακροπρόθεσμη. Άρα λοιπόν ε, παραμένει κάπως προβληματικό το θέμα. Έχουμε βέβαια ευρύτατο τύπο, ευρύτατο μάλλον φάσμα πληροφοριών και δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για κάποιες ε, συγκεκριμένες έρευνες θα πρέπει να μιλάμε για τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται και για αναλυτικούς στόχους. Η Κομισιόν πρέπει λοιπόν να δώσει απαντήσεις αλλά και το Συμβούλιο επίσης. Η Κομισιόν ίσως θα μπορούσε να αναζητήσει εναλλακτικέ λύσεις σε αυτή τη συμφωνία. Ε, ίσως τώρα, ίσως ε, σε το πλαίσιο μιας προσέγγισης σε παράλληλων οδών αργότερα, γιατί εδώ μιλάμε για την διαβίβαση στοιχείων ε, χίδιν, αν θέλετε. Δεν λύνεται το θέμα, λοιπόν, σε αυτό το, στο πλαίσιο μάλλον ετού της εδώ της εντολής. Υπάρχουν διάφορα θέματα όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία, τη δυνατότητα διόρθωσης αυτών. Ποιο είναι το σημείο εκκίνησης, ότι δηλαδή θα πρέπει ναι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι να έχουν το δικαίωμα να αναλύουν ε, στοιχεία, okay, αλλά ποια ακριβώ θα είναι τα δικαιώματα των Αμερικανών και ποια ακριβώ θα είναι τα δικαιώματα των Ευρωπαίων. Γνωρίζω πολύ καλά πω πρόκειται για μια εντολή, αλλά θέλω πολύ συγκεκριμένες απαντήσει από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν για αυτά τα πολιτικά ζητήματα που ε, μας απασχολούν. Νομίζω πως θα είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επισήμως μου είπαν ότι μπορεί να είναι και τα γενέθλιά σα σήμερα. Παρακαλώ λοιπόν να δεχτείτε τις καλύτερε ευχέ μας. Χρόνια σας πολλά. Για να ακούσουμε τώρα την Κομισιόν, τον κύριο Φόρντ. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και από την Κομισιόν προς την Ζανίν. Πολλές ευχές για τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, πρόκειται για τις απαρχές μιας διαδικασίας. Δεν πρόκειται για συμφωνία. Αυτή είναι πρόταση της Κομισιόν για διαπραγματευτικές κατευθυντήριες γραμμές από το Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει διαβουλευθεί, άρα δεν ξέρουμε και επακριβώς ποιο ακριβώς θα είναι το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ούτε βέβαια ξέρουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση αφού χρειάζονται δύο πλευρές για να διαπραγματεύονται και ακόμη με τους Αμερικανούς φίλους δεν έχουμε αρχίσει διαπραγματεύσεις και δεν θα είναι και εύκολες αυτές διότι είναι περίπλοκο το θέμα και πολιτικό και οικονομικό είναι σειρά θεμάτων Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τα μηνύματα του Κοινοβουλίου και της ε, εξαιρετικής ε, εισηγήτριας και εγκρίναμε ε, κάτι που θεωρούμε ότι είναι φιλόδοξο πλαίσιο διαπραγματευτικών κατευθυντήριων γραμμών. Οι διασφαλίσεις προστασίας δεδομένων είναι ακόμα καλύτερες από ότι εκείνες που υπήρχαν στην προηγούμενη συμφωνία που δεν την εγκρίνατε. Και ενθυμούμενοι πόσο δύσκολη ήταν η διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση εκείνης της συμφωνίας με τους Αμερικανούς, θα ήθελα να πω ότι οι διαπραγματεύσεις για την Κομισιόν θα περάσουν από δύσκολες στιγμές. Πάντως, ε, η δημοκρατική φωνή του Κοινοβουλίου έχει ακουστεί και γι' αυτό αρχίζουμε διαπραγματεύσεις ε, αποφασισμένοι να ε, παλέψουμε για μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων. Έτσι λοιπόν τα δικαιώματα για αποτελεσματική ε, διοικητική και δικαστική προσφυγή θα πρέπει να παρέχεται ε, σε βάση χωρίς διακρίσεις, δικαιώματα πρόσβασης σε διαγραφή διόρθωση δεδομένων θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία, μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία επανεξέτασης από την πλευρά μας ε, τη συμφωνίας. Θα πρέπει και αυτή να παρέχεται πέρα από τακτική υποβολή εκθέσεων από την Κομισιόν προς το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθεμάτων όπως ποσότητα, όγκος μηνυμάτων, ε, η διαδικασία TFTP, τι πληροφορίες TFTP, ε, όπου έχει χρησιμοποιηθεί ε, οι αιτήσει για δεδομένα θα πρέπει να εξετάζονται από δικαστική αρμόδια αρχή. Η νέα εντολή διευκρινίζει ότι μόνο σημαντικές πληροφορίες και όχι ε, ε, πολλά δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται για την μάχη κατά της τρομοκρατίας και θα ε, υπάρχει και ένας περιορισμός ε, σε σχέση με την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, δεν θα μπορούν να, γίνουν, να γίνονται έρευνες για δεδομένα εκτός και αν υπάρχει λόγος να υποπτευόμεθα ότι κάποιο πρόσωπο ενέχεται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να ε, τερματίσει τη συμφωνία αν υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση των διασφαλίσεων προστασίας δεδομένων. Ελπίζομαι πραγματικά ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες γρήγορα πλέον. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο στις 22 και 23 Απριλίου θα μπορέσει να εγκρίνει την εντολή. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό, αλλά ελπίζομαι και εν τη αυτή περιπτώσει θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στις αρχές Μαΐου και θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Καθ' όλη την περίοδο αυτή θα ενημερώνουμε άμεσα και πλήρως το Κοινοβούλιο για να ε, παραθέσω τη συνθήκη με τους εισηγητές, τους κοιόδης, τους συντονιστές της Επιτροπής σας ή οποιουσδήποτε άλλους ε, βουλευτές θα κρίνετε εσείς ότι πρέπει να ενημερωθούν. Ε, η διαδικασία αυτή μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων ελπίζομαι ότι θα είναι αμοιβαία και είναι σημαντική για να διασκεδαστούν οι εσδήποτε παρεξηγήσεις που έχουν ανακύψει ή που θα ανακύψουν στο μέλλον αντιλαμβανόμεθα μετά από πρόσφατες συζητήσεις ε, ε, για το SWIFT ότι τώρα έχουν κληθεί ε, στις αρχές του έτους να καταθέσουν μετέφεραν δεδομένα στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεδομένα όχι μόνο από ευρωπαϊκού σερβερ θα διατηρήσουν τα δεδομένα αυτά στους ευρωπαϊκούς σερβερ, δεδομένα τα οποία ζητήθηκαν αλλά ακόμη δεν διαβιβάστηκαν και από ό,τι αντιλαμβανόμεθα έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, για να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα και το θέμα είναι επίμαχο, ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Δηλαδή, η, αμοιβαία, ε, η συμφωνία για την αμοιβαία νομική συνδρομή είναι ο καλύτερος ή ο μόνος τρόπος οργάνωσης αυτού του συστήματος ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικά συστήματα. Επί του παρόντος ε, δεν βλέπουμε, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, κάποιο εφικτό εναλλακτικό σύστημα. Όμως ε, είμαστε ανοιχτοί στο θέμα. Προφανώς το κράτος μέλος ή τα κράτη-μέλη όπου τα δεδομένα κρατηρούνται και από το οποίο θα πρέπει να διαβιβαστούν είναι τα άμεσα ενδιαφερόμενα για το θέμα αυτό, αλλά βέβαια τίθεται ένα γενικότερο θέμα που αφορά όλο το νομικό περιβάλλον όπου όλα αυτά λαμβάνουν χώρα, οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και σίγουρα ε, θα είναι ένα σημαντικό θέμα στη συζήτηση και στο Συμβούλιο επίσης. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πραγματικά δύσκολο να δούμε κάποιο εναλλακτικό σύστημα που να λειτουργεί πέρα από αυτό. Αυτό είναι μια παραλλαγή της αμοιβαίας ε, νομικής συνδρομής και γι' αυτό ε, τόσο καιρό ε, μας πήρε να διαπραγματευτούμε και να επικυρώσουμε ένα σύστημα αμοιβαίας νομικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος να συνεχίσουμε. Η νομική βάση υφίσταται. Όμως θα εξετάσουμε και εναλλακτικέ γιατί μας ζητήθηκε αυτό και από την Προεδρία του Συμβουλίου και συνάγω από αυτά που είπατε και από εσάς και αυτό θα το κάνουμε με ανοιχτό πνεύμα. Θέλουμε ένα λειτουργικό σύστημα αποτελεσματικό που θα επιτρέπει τις απαραίτητες νομικές ε, διασφαλίσεις και βεβαίως παράλληλα τα ε, δεδομένα που θα πρέπει να διαβιβάζονται, θα διαβιβάζονται για, την, για το σκοπό της καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας. Οπότε πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές ε, αισιόδοξα, πολλά πρέπει να γίνουν. Ελπίζουμε ότι τα τρία θεσμικά όργανα της Ένωσης, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινηθούν ε, με πνεύμα συνεργασίας, παράλληλα θα υποβάλλονται εκθέσεις, θα είμαστε σε επαφή, πρέπει να αποδείξουμε ότι αντιλαμβανόμεθα πολύ καλά ότι οι διασφαλίσεις για την προστασία δεδομένων είναι περισσότερες, ισχυρότερε από ό,τι στην προηγούμενη συμφωνία. Όλα αυτά θα τα τηρήσουμε και όταν αρχίσει αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με βάση την εντολή, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια των κανόνων μας, ώστε να σας κρατούμε πάντοτε ε, πλήρως ενήμερους για τις προόδους στην διαπραγματευτική διαδικασία. Υπάρχει ένας στόχος ε, κοινός για όλους. Δηλαδή το σύστημα να έχει ε, ισχυρή νομική βάση και ένα σύστημα που θα προστατεύει αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων ε, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης της τρομοκρατίας και προς το συμφέρον το δικό μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φόλ. Και τώρα ο λόγος στα, ε, στους ε, συναδέλφους να προσθέσω κάτι στις παρατηρήσεις του κύριου Φόλ. Δεν συμφωνώ με την απόλυτη απογοήτευση που εξέφρασε η συγγήτρια. Είδαμε τεράστια πρόοδο, πιστεύω, που δεν έχει να κάνει τόσο με το κείμενο ή με τα κείμενα, αλλά αφορά κυρίως τη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αν μη τι άλλο, το όλο αυτό εγχείρημα μέχρι τώρα επιβεβαίωσε τη θέση του Κοινοβουλίου. Ελπίζω τούτο να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των επιδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Βεβαίως και βελτιώθηκε και πολύ το κείμενο που έχουμε μπροστά μας ε, τώρα. Πολλές από τις ανησυχίες που είχε εκφράσει το Κοινοβούλιο εν τέλει κάπως υιοθετήθηκαν και όπως είπε και ο κ. Φόλ βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ προκαταρκτική φάση των διαπραγματεύσεων στην ουσία εμείς ε, συζητούμε το κείμενο του εισεντολής, όχι το κείμενο αυτό καθεαυτό. Οι εισηγήτρε λοιπόν και οι σκιώδεις εισηγητέ έχουν ακόμα πολύ δυνατότητα παρέμβασης μπροστά τους και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή γιατί υπάρχει πλήρης βούληση του Κοινοβουλίου να ενημερώνεται. Να σας πω ότι το μόνο άλλο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι το θέμα του, του χρονοδιαγράμματος. Ο κ. Φολ είπε ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει την εντολή. Ελπίζω το Συμβούλιο να προχωρήσει. Είπε ότι υπάρχει, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και εσείς το είπατε κύριε Πρόεδρε στο Συμβούλιο. Εμεί αυτό το θέμα των, των ημερομηνιών πρέπει να το προχωρήσουμε και όταν υπάρχει, όσο νωρίτερα υπάρξει καλή συμφωνία, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια θα υπάρξει για τους πολίτες μας. Ελπίζω βέβαια να συνεχίσουμε να έχουμε μια κάπως διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία αυτή με άλλες όπως το SWIFT και το PNR. Ανέφερε ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ναι μεν υπάρχουν ομοιότητες σε ό,τι αφορά την παροχή δεδομένων, αλλά ότι τα θέματα αυτά είναι διαφορετικά και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και μέσα στο δικό τους χρονοδιάγραμμα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να εμπλέξουμε τις δύο αυτές τα δύο αυτά νομικά κείμενα στην ευρύτερη, στη, στις ευρύτερες σχέσεις ένωσης ΕΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι τα θέματα που αντιμετωπίζουμε έχουν εμπολίσει καλυφθεί και ελπίζω να υπάρχει μια ικανοποιητική, να υπάρξει γρήγορα μια ικανοποιητική λύση στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, όπως ακούσατε, στην εντολή υπάρχουν ορισμένα θέματα που δεν βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο το Κοινοβούλιο. Παράδειγμα, εξατομίκευση της διαβίβευσης αντί γενική διαβίβαση δεδομένων. Ε, δηλαδή, δεν πρόκειται για αρχή, αλλά για δικαστή που θα πρέπει να αποφασίσει για τη διαβίβαση ποιων δεδομένων. Επίσης, ε, μπαίνει θέμα ασφάλειας δικαίου και για τις ΗΠΑ Πολιτείες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η διάρκεια της αποθήκευσης 5 έτη είναι υπερβολικό το διάστημα αυτό. Θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται αυτό στις αρχές ε, προστασίας δεδομένων και εμείς ακόμα δεν έχουμε αποδείξει στοιχεία για την ε, αναγκαιότητα της διαβίβασης αυτών των τραπεζικών δεδομένων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Βέβαια, κάποια αποδεικτικά στοιχεία έχουν υποβληθεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τελεσίδικα. Δεν μας πείθουν δηλαδή ε, σε σχέση με την αναγκαιότητα ε, στα πλαίσια του TFTP. Άρα λοιπόν μπαίνει ένα θεμελιώδες ερώτημα της ανάγκης για αυτά τα στοιχεία. Γιατί αυτό είναι το καθοριστικό. Εάν θέλω να κρίνω την αναλογικότητα των μέτρων και το κατά πόσον υπησέρχονται στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών. Ε, άλλωστε, αυτή η κριτική δεν γίνεται μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια κριτική που αφορά συγκεκριμένα σημεία, πρόκειται για προϋποθέσεις πλαίσιο που έχουν επιβληθεί, αν θέλετε, ε, από εμάς σε συνταγματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές συμβάσεις ε, στα άρθρα 6, 13 ε, υπάρχουν ε, ορισμένες διασφαλίσεις προστασία δεδομένων και δεν διασφαλίζονται από ό,τι βλέπω από την εντολή 100%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξακολουθήσουν οι εργασίες πάνω στο θέμα αυτό. Εδώ και περίπου τέσσερις μήνες αυτά τα δικαιώματα υπάρχουν και στο θεμελιώδη ε, χάρτη. Και αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα σε σχέση με την κατάσταση πέρυσι. Άλλωστε θα πρέπει να δούμε ότι αυτό έχει και ε, ουσιαστικές επιπτώσεις. Υπάρχουν δηλαδή και αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Γερμανία για την αποθήκευση των δεδομένων. Γιατί όταν χρησιμοποιούμε ε, τέτοια δεδομένα, το Συνταγματικό Δικαστήριο θέτει ε, ε, μεγάλους φραγμούς εις ό,τι αφορά τη χρήση των δεδομένων. Και υπάρχει ο κίνδυνος, για παράδειγμα, η Γερμανία να αναγκαστεί να απορρίψει την εντολή εάν θέλει να σεβαστεί τις, τις αποφάσεις του δικού της συνταγματικού δικαστηρίου. Υπάρχουν συνταγματικοί φραγμοί και εμπόδια. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν εσείς ως Κομισιόν να κάνετε ένα βήμα μπροστά ούτω ώστε να ε, βελτιώσετε τα ε, θέματα αυτά που αφορούν τα συνταγματικά εμπόδια επί των οποίων δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουν εντατικά οι εργασίες πάνω στην εντολή. Ευχαριστώ. Κύριος Λαμπρινίδης. Ευχαριστώ. Κατά το παρελθόν Είχαμε πολλές ανησυχίες σημαντικές ισότι; αφορά την ε, πολιτική των ΗΠΑ κατά τις διαπραγματεύσεις των θεμάτων αυτών. Και βεβαίως είχαμε και κάποια θέματα εις ό,τι αφορά την ικανότητα της δικής μας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κρατήσει στεναρή στάση. Πρέπει να πω μετά τα αρχικά σχόλιά σας σχετικά με τις δυσκολίες κατά τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η αίσθησή μου μετά από ε, συνομιλίες που είχα για το θέμα στο πρόσφατο παρελθόν είναι ότι υπάρχει καλή θέληση από την Αμερικανική κυβέρνηση τώρα ε, σε, και αυτό διαφοροποιεί πολύ την κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν στις διαπραγματεύσεις, ε, εάν παρουσιάσετε έγκυρα επιχειρήματα ε, και τα παρουσιάσετε στεναρά, ε, θα αντιμετωπιστούν με καλύτερο τρόπο. Στις διαφορές θα σας στηρίξει το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να επιληθούν τα θέματα προς, το, προς την κατεύθυνση της άποψης του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω, τώρα, τρεις ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Δεν ξέρω αν το είπε πολύ κτενός η Ζανίν. Ε, τι γίνεται με την ε, διαβίβαση ε, μεγάλων όγκων δεδομένων. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να πάρουμε μερικά δεδομένα πέραν αυτού, δηλαδή με μεγάλο όγκο διαβίβασης. Το SWIFT ισχύει ότι δεν μπορεί να απομονώσει δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως λέτε, ή απλώς δεν το κάνουν, αρνούνται να το κάνουν. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι τεχνικό ή λόγω της εταιρική τους ε, κουλτούρας δεν θέλουν να συνεργαστούν πάνω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αν συνεχίζουν να στέλνονται αυτά τα χίδινα αν θέλετε, δεδομένα, πρέπει να δούμε τα εξής και να τα απαντήσουμε. Πρώτον, τι διασφαλίσεις έχουμε κατά νου για να προτείνουμε στους Αμερικανούς τις διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσουμε έτσι ότι αυτή η μεγάλη διαβίβαση δεν θα ε, οδηγεί σε παραβιάσεις. Το SWIFT σήμερα έχει διασφαλίσεις δικές του που έχει διαπραγματευτεί με την έγκριση των ΗΠΑ. Θα διατηρηθούν, θα βελτιωθούν αυτές. Δεύτερον, ε, με τη διπλή προσέγγιση της Ρανίν έχει σχέση αυτό. Γιατί να μην σκεφτούμε έναν τρόπο, είτε για το ίδιο το SWIFT, ή για κάποια άλλο ευρωπαϊκό οργανισμό για να γίνεται η αναζήτηση που θέλουν οι Αμερικανοί και να σταματήσουμε να τους στέλνουμε αυτά τα χίδιν ε, μηνύματα και στοιχεία. Επίσης το SWIFT εξακολουθεί να έχει σερβερ ε, νόμιζα τον είχαν κλείσει και ε, μετέφεραν όλα στην Ευρώπη. Τι δεδομένα τηρούνται σε αυτό το σερβερ και τι όχι. Επίσης, τρίτο ερώτημα που αφορά τις τρίτες χώρες που ε, αναφέρατε και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Είναι καλό που η συμφωνία όπως την περιγράψατε θα περιορίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που θα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Όμως μέχρι σήμερα δεν είναι καλό το γεγονός ότι δεν υπάρχει απέτηση από τις ΗΠΑ να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όντως διαβιβάζει τέτοια στοιχεία σε τρίτες χώρες. Το ίδιο πρόβλημα το είχαμε με τη Συμφωνία PNR. Ε, θέλαμε να διαπραγματευτούμε πολύ, και ήταν πολύ αυστηρά τα ε, ε, πολύ ε, αυστηρές οι ε, προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση ε, των δεδομένων τους προς εμάς, αλλά ήταν πολύ πιο γενναιόδορη και χαλαρή σε ό,τι αφορά ε, τη μεταφορά, τη διαβίβαση δεδομένων δικών μας προς τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει απέτηση οι διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες των δεδομένων να εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν προχωρήσουν στη διαβίβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια τεχνική παρατήρηση. Δεν λειτουργούν τα ακουστικά μας. Ας τα ελέγξουν οι τεχνικοί γιατί έπρεπε να δανείζομαι τα ακουστικά του κυρίου Βέμπερ. Τώρα, επί της ουσίας. Συμφωνώ με εκείνους που λέγουν ότι είπα θέλουν να διαπραγματευτούν και αυτό είναι θετικό. Παράλληλα έχει δίκιο και ο κύριος Φόλ που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι απλές βεβαίως. Ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι καλά θα κάναμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ στεναροί στις θέσεις μας κατά τις διαπραγματεύσεις, γιατί όποιος πάει στις διαπραγματεύσεις με συμβιβαστικό πνεύμα ευθύ εξ αρχή θα καταφέρει πολύ λιγότερα από ότι αν θέσει αιτήματα ευθύ εξ αρχή. Γι' αυτό συμφωνώ και με την κυρία Πλέσσερτ που είπε ότι ε, πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο το σχέδιο της εντολής. Μας απογοητεύει σε ορισμένες πτυχές, δεν διευκρινίζει κάποια θέματα. Επίσης, αμφιβάλλω αν ε, η SWIFT από τεχνικής άποψης είναι σε θέση να ξεδιαλέγει τα δεδομένα, να τα επιλέγει κάθε τράπεζα μπορεί συγκεκριμένα δεδομένα από συγκεκριμένα πρόσωπα να τα ξεδιαλέγει. Δεν μπορεί να είναι μεγάλο το τεχνικό <laughs> πρόβλημα μια εταιρεία όπως η SWIFT να μην μπορεί να το κάνει και να στέλνει σοριδών τα δεδομένα στις ΕΠΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ε, θέμα κέριο στην κριτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι ένα πράγμα πρέπει να διευκρινίσουμε. αν το τέλος των διαπραγματεύσεων η συμφωνία δεν διαφοροποιείται πολύ από αυτή που απορρίψαμε, ε, δεν μπορούμε και να την εγκρίνουμε, γιατί θα γελιοποιηθούμε. Εάν απορρίψουμε μια συμφωνία με σοβαρά επιχειρήματα και μετά, επειδή έχουν γίνει μικροαλλαγές, να το δεχτούμε είναι σαφές ακόμα το θέμα της διαβίβασης των δεδομένων, δηλαδή όλα μας τα δεδομένα θα πρέπει να διαβιβάζουμε στις ΕΠΑ. Δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί και δυνατότητες διαλογής. Δεύτερον, όταν πρόκειται για μεμονωμένα πρόσωπα και αυτό το ρώτησα στο Υπουργείο Οικονομικών όταν πρόκειται για συγκεκριμένα δεδομένα μεμονωμένων προσώπων ή οργανισμών αν πρόκειται γι' αυτό τότε ε, έχουμε την ε, αμοιβαία συνδρομή οι Ηνωμένε Πολιτείε συμφωνούν με αυτό. Λένε ναι, λειτουργεί το σύστημα σε αυτέ τι περιπτώσει, παρόλο που παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο. Αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα όπω το SWIFT, πρέπει να υποθέσω ότι δεν πρόκειται μόνο για το φιλτράρισμα συγκεκριμένων προσώπων. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να διευκρινιστεί. Το θέμα του χρόνου ε, φύλαξης των δεδομένων, αν χρειάζομαι από χιλιάδες δεδομένα μόνο τρία, όλα τα άλλα θα φυλάσσονται για πέντε χρόνια. Για ποιο σκοπό. Και αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, για οδήποτε σκοπό, για ε, ε, ούτως ώστε μέσα στην πενταετία να μπορεί να ε, έχει κανείς πρόσβαση στα αυτά τα δεδομένα ή υπάρχουν άλλοι λόγοι. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και η διαβίβαση σε, τρίτα, σε τρίτες χώρες και αυτό είναι προβληματικό. Μπορεί να πρόκειται για κάποιον ύποπτο για τρομοκρατική δραστηριότητα. Ε, πάλι η διαβίβαση δεδομένων δεν πρέπει να γίνονται σε όλες τις χώρες αδιακρίτως και εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί στην εντολή αν μπορεί να υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί. Και το θέμα της ασφάλειας δικαίου και τι δυνατότητες υπάρχουν και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί. Πιο σημαντικό είναι το θέμα ε, της διαβίβασης λιγότερων δεδομένων γιατί έτσι η ασφάλεια δικαίου θα υποφέρει ε, λιγότερο από ότι αν ε, διαβιβάζουμε ε, τα δεδομένα μας. Η κυρία Ινφέλτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επειδή υπόθηκαν όλα από όλου, επαναλάβω ορισμένα από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι, αλλά με διαφορετική διατύπωση. Και έχοντα υπόψη βέβαια και την ανάγκη να συμπεράσματα που θα έχουν αντίκτυπο για τι συζητήσει για το PNR παρότι πρόκειται για διαφορετικό θέμα και συμφωνώ με τον κύριο Κίρκοπ. Αυτά που είπε και η κυρία Σίπελ, το βασικό θέμα είναι το θέμα της, απλο... αναλογικότητας. Με λίγα λόγια, οι Αμερικάνοι ψάχνουν μία βελόνα και εμείς του στέλνουμε ένα ολόκληρο κουτί με άχυρα. Αυτό είναι το θέμα. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι μόνο Ηνωμένε Πολιτείε. Δείτε και την κατάσταση του PNR. Όλο και περισσότερε χώρε, όχι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε, όχι μόνο Καναδά, η Αυστραλία, η Κορέα, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, θα ζητούν στοιχεία PNR. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα υπάρξουν οι ίδιε εξελίξει και στα οικονομικά, χρηματοοικονομικά, χρηματοπιστωτικά δεδομένα. Άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε προηγούμενο. Εμεί πιστεύουμε πάντα ότι το φιλτράρισμα των δεδομένων, η προσπάθεια να βγάλουμε τη βελόνα, δεν ήταν τεχνικά δυνατό. Γι' αυτό στείλαμε ολόκληρο το φορτίο με τα άχυρα. Αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι το θέμα είναι θέμα χρημάτων. Το SWIFT λέει δεν δική μας δουλειά. Σωστό. Λένε είναι ακριβό. Πιστεύω ότι το φιλτράρισμα θα πρέπει να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα αρχής που θα πρέπει να αφορά όλα τα θέματα διαβίβασης δεδομένων, χρηματοπιστωτικά, PNR, δεδομένα τηλεπικοινωνιών, οτιδήποτε. Διότι είναι ένα ζήτημα, όχι ίδιο, αλλά συ, συγκρίσιμο. Τι κάνουμε στο push and pull, τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπαίνουν στα δικά μας συστήματα κρατήσεων στα κομπιούτερ των συστημάτων κράτησης. Οι Αμερικανοί θα κάνουν το ίδιο με εμά. Δεν το πιστεύω. Και πολύ σωστά δι, αρνούνται να μας δώσουν το, το, login. Και εμεί το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Διαπραγματεύσεις τώρα. Όντως θα είναι δύσκολες. Γιατί το λέμε όμως συνέχεια. Ότι στην περίπτωση αυτή ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αυτές που ζητούν από εμά. Γιατί εμείς ξεκινούμε λέγοντας ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Η δουλειά μας είναι να προσπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας και να έχουμε καλές σχέσεις με τους φίλους και, και εταίρους. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ε, να λέμε ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Το θέμα της αναλογικότητας θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις ε, διαπραγματευτικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που τώρα μόλις ξεκινά στην Ευρώπη. Η συζήτηση για την προστασία των δεδομένων ξεκινά Δυστυχώ να συνδέεται όχι μόνο με την τρομοκρατία, αλλά και με το οργανωμένο έγκλημα την ε, διεθνή τρομοκρατία, ε, τη, διεθνή εγκληματικότητα. Είναι λοιπόν μια συζήτηση που θα συνεχιστεί. Είναι γεγονό ότι με την νέα εντολή μπαίνουμε σε κάποια ζητήματα ουσία. Θα πρέπει ωστόσο να συνεχίσουμε να δουλεύουμε τα θέματα αυτά, διότι κάτι τέτοιο δεν συνδέεται με τα PNR. Υπάρχουν πολλά συστήματα που δημιουργούν άρση εγγύσεων και όχι μόνο αυτά που συζητούμε και αναλύουμε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι η συζήτηση είναι μεγάλη και ξεκινά. Επίσης πρέπει να είμαστε να συνδυάζουμε τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει ε, ασφάλεια. Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη χώρες που έχουν περάσει η τρομοκρατία μαζικά και χώρες που δεν έχουν μαζικές επιθέσεις τρομοκρατικές, ε, τρομοκρατικού χαρακτήρα. Αυτές δημιουργούν πανικό στον πληθυσμό. Και όταν υπάρχει πανικός στον πληθυσμό, οι κυβερνήσεις δρούν με δυσανάλογο τρόπο, σε πολλές περιπτώσεις με τη συνένεση των πολιτών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς και προγράμματα όταν δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα να το κάνουμε. Πιστεύω ότι το πρόβλημα, το αρχικό πρόβλημα, είναι ένα πρόγραμμα ε, μαζικό. Και εφόσον είναι μαζικό, είναι δυσανάλογο. Στην περίπτωση ε, των Ηνωμένων Πολιτειών η αντιμετώπιση αυτή ξεκίνησε μετά την επίθεση στους Δήμους Πύργους. Αυτό που είναι παράλογο είναι αυτό το, το σύστημα ε, μαζικών περιορισμών και άσεων των εγγύσεων δεν πρέπει να κρατά επιμακρών. Διότι όταν δεν ήταν αυτό το σύστημα αποτελεσματικό τότε τι νόημα έχει να γίνει σήμερα η Αμερική ο παγκόσμιο χωροφύλακα που θα εξετάζει όλε τι τρομοκρατικέ δραστηριότητε στον κόσμο. Δεν μπορούμε εμεί να υλοποιούμε τα δικά μα μέτρα όταν έχουμε τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε τα δικά μα συστήματα πρόληψη. Δεν είμαστε εμεί ικανοί να ε, υιοθετήσουμε συστήματα που θα έχουν αναλογικότητα σε σχέση με την απειλή. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όταν λοιπόν λέμε ότι η ίδια εταιρεία SWIFT θα είναι αυτή που θα επιλέγει τα στοιχεία. Λάθος. Μηνύματα στέλνει. Δεν έχει ούτε δικαστικό ούτε αστυνομικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι αδύνατο να το κάνει η επιχείρηση αυτή. Είναι μια επιχείρηση που κάνει data messaging. Αυτή είναι η δουλειά της. Πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη συζήτηση και θα έπρεπε να εξετάσουμε ένα κατά πόσον το πρόγραμμα ή το εργαλείο που δημιουργείται είναι αναλογικό για να προστατεύονται τα δεδομένα, προφανώ. Επιπλέον δε, τι πλαίσιο να ζητούμε για να είμαστε σε θέση να προλαμβάνουμε μία απειλή. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας, στη συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Δυστυχώς αυτά τα συστήματα είναι συστήματα προληπτικά. Το ξέρει ο κύριος Φολ. Μιλάμε για πρόληψη της δημοκρατίας Άρα μιλούμε για έρευνα υπόπτων, σε ύποπτους. Σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία αυτή δεν έχει μπει στο δικαστικό πλαίσιο. Το να μπαίνει λοιπόν μια επιχείρηση να κάνει αυτή τη δουλειά με, με φοβίζει. Θα τόνιζα λοιπόν ότι ίσως θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ε, μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος. Διότι οι επιχειρήσεις ε, αποστολής δεδομένων δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία αυτή όπως θα έπρεπε. Αν ήταν μέσα στην οδηγία ως υπόχρεοι θα είχαν την υποχρέωση να προσφέρουν πληροφορίες. Ωστόσο οι πληροφορίες που δίνουν πρέπει να θεσπίσουμε σε ποιο πλαίσιο θα δίνονται. Διότι στους υπόλοιπους υπόχρεους το πλαίσιο θεσπίζεται. Και εκεί μπορούμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα. Όταν μπαίνουμε σε ένα, φτάνουμε σε ένα αεροδρόμιο πρέπει να δηλώσουμε. Έχουμε πάνω από 10.000 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο είναι το ποσό, αν έχεις μαζί σου πάνω από 10.000 ευρώ πρέπει να τα δικαιολογήσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της μάχης κατά της, ε, του ξεπλήματος κεφαλαίων που είναι χρηματοδότηση της δημοκρατίας και που είναι η βάση, η ουσία βάση της συμφωνίας αυτής, πρέπει να υπάρξει μια διεθνή συνεργασία σε πολύ πιο ομοιογενή βάση. Στις ομάδες χρηματοοικονομικής, στην ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης συζητούν αυτή την ε, τυποποίηση, την, ε, την ομοιομορφία των προτύπων. Και εκεί θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς την οδηγία μας για να συμπεριλάβουμε ε, τέτοιες επιχειρήσεις. Επιπλέον ωστόσο, Πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι αρκετά κάθε, αρκετό κάθε κράτος μέλος να προχωράει μόνο του. Εμείς στην Ισπανία προχωρήσαμε γιατί είχαμε σφαγές λόγω τρομοκρατίας και προχωρήσαμε με βάση την οδηγία ξέπλυματος των κεφαλών όπου αντιμετωπίζονται ζητήματα προστασία ε, προστασίας δεδομένων, ε, παρουσίας της ε, δικαιοσύνης, ε, αστυνομικής Ωστόσο, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός που να κάνει το ίδιο πράγμα που κάνουμε εμείς σε εθνικό επίπεδο σε ευρωπαϊκό. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένα εργαλείο αμοιβαιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ήταν ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με το Ηνωμένων Πολιτειών που είναι μπαίνουμε παντού είναι λάθος. Δεν έχουμε σήμερα μια απειλή παρόμοια. Η ευθύνη που έχουμε ως κοινοβούλιο είναι να μπορέσουμε να μετρήσουμε την απειλή σε σχέση με την αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Κύριε Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚΟ, ο Στράσερ, δεν μπορούσε να έρθει και τον αντικαθιστώ. Καταρχήν τα θετικά. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι Έχουμε μάθει το μάθημά μας μετά από αυτά που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Οπότε καλωσορίζομαι το γεγονός ότι η Κομισιόν είναι πιο ανοιχτή, πιο πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί μας σε θεσμικό επίπεδο. Επίσης εκτιμούμε το γεγονός ότι η Επίτροπος Μάλμστρομ ήρθε αμέσως σε μας μετά την έγκριση του, της διαπραγματευτικής εντολής από την Κομισιόν και αυτό είναι καλό. Το δεύτερο θετικό είναι ότι γενικά πιστεύουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο ε, και επί της ουσίας ε, και εκτιμούμε την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλών παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα εκεί όπου επέμεινε στο ψήφισμα. Βέβαια, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως λένε. Και εδώ περνάμε πια στην πραγματική πολιτική αντιπαράθεση όπου ως θεσμικό όργανο θέλουμε να υπάρξει κάποια διαφορά στην έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων κύριε Φόλ και εδώ συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν ο κύριος Λαμπρινίδης, η κυρία Σόφη Ίντφελτ και άλλοι σε ό,τι αφορά την ε, σοριδόν διαβίβαση δεδομένων. Δεν μιλάμε εδώ για περιορισμό των ομαδικών αποστολών ή την ομαδική διαβίβαση. Θέλουμε να αποφεύγονται οι ομαδικές διαβιβάσεις γενικώ. Καταρχήν. Και υπάρχει εδώ ε, ένα ποιοτικό άλμα ε, σε αυτό που ισχυρίζεται το θεσμικό μας όργανο. Δηλαδή, είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το ερώτημα θέτω προς την Κομισιόν, γιατί για μας αυτό το θέμα είναι κέριο. Βέβαια θα ήταν πολύ πιο καλό οι Αμερικανικές αρχές να έχουν μια ε, συνεργασία με τη Europol για παράδειγμα όταν πρόκειται για θέματα ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών παρά οι Αμερικανικές αρχές να συναλλάσσονται άμεσα απευθείας με τη SWIFT εις ό,τι αφορά τις πληροφορίες που φυλάσσονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οπότε αυτό είναι ένα κύριο ζήτημα και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Επίσης το θέμα της προσφυγής. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι μέχρι τώρα. Ειδικότερα, τι δικαιώματα έχει το πρόσωπο που νιώθει ότι προσβάλλεται από τις πληροφορίες που φυλάσσονται γι' αυτόν, αν τα δικαιώματα του προσώπου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που έχουν οι Αμερικανοί ε, εταίροι μας, οι ομολογοί μας. Βεβαίως, ο χρόνος είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Θέλουμε συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν, αλλά είναι σαφές από τη συζήτηση αυτή ότι δεν θέλουμε συμφωνία ε, με κάθε τίμημα και βέβαια ε, θέλουμε να στηρίξουμε την, εισηγή, την εισηγήτρια, θέλουμε να αναδειχθεί αυτό. Πιστεύουμε ότι η δική της γραμμή πλεύσης είναι η σωστή και η ακολουθητέα. Τέλος, η αξιοπιστία της Κομισιόν διακυβεύεται εδώ. Η Κομισιόν έχει μεγάλη ευθύνη στις διαπραγματεύσεις αυτές, ώστε να διασφαλίσει ότι θα διαχειριστεί ένα αποτέλεσμα καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα πλαίσια των διεθνών διαπραγματεύσεων. Ε, αυτή την έννοια θέλω να διευκρινίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα η Επιτροπή μας θα ακολουθήσει μια επικοδομητική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ. Πριν επανέλθουμε στην εισηγήτρια την κυρία Χένις Πλάσερτ, ίσως η Προεδρία ε, θα μπορούσε να μας πει... Θέλει το λόγο στη συζήτηση αυτή. Κύριε Αγγιλέρα. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση. Οι συμπληρωματικέ πληροφορίες που θα μπορούσα να σας ε, δώσω τώρα είναι ότι είχαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο το Φεβρουάριο, στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου μια πλειοψηφία κρατών μελών συμφώνησαν για την σκοπιμότητα του να προχωρήσουμε στην σύναψη μιας νέας συμφωνίας εντάχει και στο νέο αυτό πλαίσιο που έχουμε και που είναι ένας στόχος που θα πρέπει να επιτευχθεί με πλήρη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή η σύσταση για το ξεκίνημα της διαπραγματεύσης που ενέκρινε τη, στις 24 Μαρτίου η Επιτροπή ε, επιτρέπει το ξεκίνημα της διαδικασία για την έγκριση ε, της εντολής στο Συμβούλιο και ξεκινά από την σύσταση της Επιτροπής ότι εν γέννη αναφέρθηκε και με την επιφύλαξη των προβλημάτων που αναφέρθηκαν και που καταγράφονται περιλαμβάνονται σημαντικές βελτιώσεις και η γενική εντύπωση που υπάρχει είναι ότι λαμβάνονται υπόψη πολλές από τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από το Κοινοβούλιο, όπως επίσης αναφέρθηκε. Θα προχωρήσουμε με ταχύτητα πρόεδρε, σε συνεργασία και ακούγοντας απόλυτα αυτά που ακούστηκαν εδώ, τις θέσεις δηλαδή που συνεχίζει να έχει το Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον στόχο, όπως αναφέρθηκε ωστόσο. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να σέβεται εγγυήσεις και να, είναι αποτέλεσμα, να έχει εν τέλει ένα αποτέλεσμα αποτελεσματικό για όλους. Αυτά προς το παρόν. Όπως ήδη σας είπα και πιστεύω ότι ε, σημαντικό. Έχουμε, ακούμε απόλυτα και προσέχουμε απόλυτα αυτά που τονίζει και θέτει το Κοινοβούλιο. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της διαπραγμάτευσης. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Κλείνουμε την ανταλλαγή απόψεων με την ε, ολοκληρή συζήτηση από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Να υποχρεωμήσω μόνο την ανάγκη να διαφοροποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ βασικών αποφάσεων πολιτικής που θα αποφασίζει η Ένωση, το Συμβούλιο, και της εφαρμογής των προβλεπόμενων συμφωνιών ΗΠΑ Ένωσης. Τονίζαν, τόνισαν όλοι οι συνάδελφοι την σημασία της αναλογικότητας. Η σοριδόν μεταφορά δεδομένων δεν μπορεί να παραμερίσει την προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων. Και με την νέα εντολή ακόμα, εγώ θεωρώ θετικό το ότι η εντολή καλύπτει μια σειρά ερωτημάτων που είχαμε θέσει, αλλά και με τη νέα εντολή μιλάμε για 90 εκατομμύρια δεδομένα μήνα. Αυτό δεν είναι εξατομικευμένα, αλλά σοριδών. Θα πρέπει λοιπόν μεταφορά δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε σαφώ στο Συμβούλιο και το Επιτροπή τι περιμένουμε στην διαπραγμάτευση. Το θέμα της μεταφοράς δεδομένων σωριδών είναι εξαιρετικά σύνθετο. Συνεχίσουμε να μεταφέρουμε την αντιτομοκρατική μας πολιτική σε μια ξένη δύναμη. Αυτό θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα. Εγώ είμαι επικοδομητική. Δεν έχουμε χρόνο, το ξέρω. Ε, πιστεύω ωστόσο ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γνωριθεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες. Πάλι δεν έλαβα απάντηση για το ότι τώρα οι πολίτες της Ένωσης θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Αμερικανούς πολίτες ή όχι. Ποια είναι όμως αυτά τα δικαιώματα σε μια τέτοια περίπτωση τι δικαιώματα θα έχουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί προφανώ πολίτε. αν η συμφωνία αυτή ε, θέλει να εξασφαλίσει αποτελεσματική προσφυγή, μη διάκριση λόγω εθνική εθνικής καταγωγής κλπ. Υπάρχει κάποιο κείμενο που λέει ποια, είναι αυτά τα δικαιώματα. Ρητά. Ευχαριστώ. Κύριε Φόλ. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτά τα σχόλια και τι ερωτήσει. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα όσο γίνεται πιο σύντομα. Βεβαίω, με την επιφύλαξη ότι οι οριστικέ απαντήσεις δεν θα είναι γνωστές μέχρι ότου να έχουμε εντολή και να έχουμε επιτυχώς ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει και να έχετε μπροστά σα μια συμφωνία επί τη οποία θα ερωτηθείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Δεν μπορώ να προβλέψω δηλαδή όλες, όλα τα ενδεχόμενα σε το στάδιο αυτό. Μια δεύτερη γενική παρατήρηση. Φυσικά θα συζητήσουμε στο Συμβούλιο και στις διαπραγματεύσεις ε, όλα ε, τα θέματα που εσείς ε, θίξατε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να σας φέρουμε μια συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα Ε, ελπίζοντας ότι θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας γνωρίζοντας και όλες τις ανησυχίες σας αλλά και τις θεμελιώδεις σας θέσεις. Φυσικά πρόκειται για νέες διαπραγματεύσεις με βάση μια νέα συνθήκη και υπάρχουν διάφορες διαφορές. Ελπίζω πως ο Σταύρος Λαβρινίδης θα έχει δίκιο ότι η καλή θέληση της Αμερικανικής κυβέρνησης θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι παλαιότερα. Ας ελπίσουμε. Πάντως από την πλευρά μας είναι νέα η κατάσταση από δύο πλευρέ. Καταρχήν η Κομισιόν θα διαπραγματευτεί εκ μέρου τη Κομισιόν. Αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Δεν θέλω να ελαχιστοποιήσω το σύστημά μα, αλλά ήταν μια ε, συμφωνία του Συμβουλίου στην οποία δεν δώσατε τη σύμφωνη σα γνώμη και σύμφωνα με τι ισχύουσε ε, συνθήκε παλαιότερα το Συμβούλιο διαπραγματευόταν ενώ η Κομισιόν ε, το υποβοηθούσε. Βέβαια δεν το λέω αυτό για να νύψω τη γύρα μου, α, κάναμε, δέχομαι τα όσα κάναμε, αλλά τώρα εμείς είμαστε επικεφαλής. Τώρα έχουμε και νέα κομισιόν και η κομισιόν αυτή πολύ σαφώς άκουσε τα όσα της είπατε στα πρώιμα στάδια της ζωής της. Δεύτερον, και εσείς συμμετέχετε με έναν τρόπο που παλαιότερα δεν ίσχυε. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε πλήρως και άμεσα και τέλος δίνετε τη συγκατάθεσή σας ή όχι. Και εφόσον αυτό το γνωρίζουμε και εφόσον θα ερχόμαστε εδώ τακτικά σε όλα τα επίπεδα ώστε να σας ενημερώνουμε πλήρως, θα λαμβάνουμε υπόψη ακόμη περισσότερο από ό,τι παλιότερα την θέση του Κοινοβουλίου. Η επιρροή σας λοιπόν σε όλη τη διαδικασία είναι τεράστια Ακόμα και αν στο τέλος της ημέρας εσείς είστε αυτοί που θα αποφασίσετε. Και θα ήταν ανόητο εκ μέρους μας να σας παρουσιάσουμε μια συμφωνία χωρίς μια κάποια ε, προηγούμενη εμπιστοσύνη ότι θα τη δεχτείτε. Σας είπα ότι τα διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες, αναμφίβολα θα είναι δύσκολες και για τις δύο πλευρές και ελπίζουμε ότι θα αξίζουμε στο τέλος να διαπραγματεύσεων της εμπιστοσύνη σας. Τελευταία γενική παρατήρηση πριν να φτάσω στις πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Και δεν το λέω αυτό έτσι ε, με οποιαδήποτε διάθεση αντιπαράθεσης. Δεν κάνουμε outsourcing στην πολιτική κατά της ε, τρομοκρατίας. Οι αντιτρομοκρατικές δράσεις είναι παγκόσμιες εμβέλειες πλέον. Κάνουμε διάφορα πράγματα για εμάς. Είναι αλήθεια πως δεν έχουμε ακόμα σύστημα PNR, το έχουμε προτείνει. Είναι αλήθεια πως δεν έχουμε τι Ναι, το, το 11 Σεπτεμβρίου έγινε στις ΗΠΑ και όχι εδώ, αλλά είναι επίσης αλήθεια πως η 11 Σεπτεμβρίου σκότωσε ένα σωρό Ευρωπαίους και ότι πολλές από τις χώρες μας έχουν πρόσφετες άμεσες τραγικές εμπειρίες τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως μας θύμισαν οι συνάδελφοι πριν από λίγο. Νομίζω, νομίζω λοιπόν πως δεν είναι δίκαιο να μιλάμε για outsourcing, ότι αναθέτουμε δηλαδή σε εξωτερικό συνεργάτη στην αντιτρομοκρατική μας δράση. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι όπως είναι. Οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει ένα σωρό ε, στοιχεία. Οι πληροφορίες είναι βεβαίως η βάση εργασίας πολλών αντιδημοκρατικων δράσεων και αστυνομικών δράσεων και άρα είναι ένα πολύ κεντρικό ζήτημα στην ε, πολιτική κατά της τρομοκρατίας ή συγκέντρωση στοιχείων και ανταλλαγή στοιχείων. Τώρα, για τον κύριο Άλμπρεχτ, η πενταετής περίοδος αποθήκευσης είναι αυτό το οποίο εμείς ε, ανασύραμε από την οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος. Ε, είναι, πιστεύουμε, ένα λογικό όριο με βάση τα όσα γνωρίζουμε σε σχέση με την ηλικία κατά την οποία οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι χρήσιμες για πιθανές έρευνες κατά της θερμοκρατίας. Αλλά τα ακούσαμε αυτό που μας είπατε και θα το πω και σε σχέση με άλλα θέματα, ότι σίγουρα θα διαπραγματευτούμε όσο γίνεται πιο σταθερά, ώστε να περιορίσουμε στο μίνιμουμ πολλά από αυτά τα θέματα. Φυσικά και γνωρίζουμε υπό ποια νομοθεσία λειτουργούμε, γνωρίζουμε τις αποφάσεις του δικαστηρίου τι αποφάσει των εθνικών δικαστηρίων και είμαι βέβαιος ότι στο τέλος όταν θα έχουμε διαπραγματευτεί μια συμφωνία στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο θα συμφωνεί πως θα, ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας στείλει προς δική σας έγκριση θα το πράξουμε μόνο εφόσον είμαστε βέβαιοι πως συμμορφούνται πλήρως με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ισχύουσες νομοθεσίες. Ελπίζω πως αυτό είναι αυτονόητο. Για τον Σταύρο Λαμπρινίδη είπατε για καλή βούληση από τη ΣΥΠΑ. Ας το ελπίσουμε. Εμείς είμαστε πιο, το Κοινοβούλιο είναι πιο ισχυρό από ό,τι παλιότερα στο ρόλο του. Εμείς είμαστε ε, βασικός διαπραγματευτής και πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις με φρέσκες ιδέες για το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε και γνωρίζοντας πως τα γεγονότα εδώ στο σώμα εισακούστηκαν και έγιναν κατανοητά, ελπίζω, και στην Ουάσιγκτον. Το θέμα των ε, μαζικών μεταφορών στοιχείων και αυτό προέκυψε σε διάφορες παρεμβάσεις, φυσικά είναι δύσκολο. Αναμφίβολα, θα ήταν καλό να, καλύτερο να έχουμε ένα σύστημα όπου θα έλεγε ε, ότι μας ενδιαφέρουν τα τάδε στοιχεία για συγκεκριμένα άτομα και θέλουμε εκείνη εκεί την βελόνα στα άχυρα, όπου και βρίσκεται. Βέβαια, το σύστημα όπως είναι τώρα σχεδιασμένο και όταν λέω το σύστημα εννοώ τόσο τις ε, λειτουργικότητες του SWIFT όσο και το πρόγραμμα κατά πολέμηση τρομοκρατίας δεν προβλέπουν τέτοιο είδους ανέβρεση βελόνας. Υπάρχει λοιπόν το στοιχείο του βουνό άχυρο, Όπως υπάρχει και το στοιχείο της μεταφοράς στοιχείων σε κάποια μεγάλο όγκο, μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια τον όγκο αυτόν και μπορούμε να δούμε και ποιο θα είναι το, ο όγκος αυτός των πληροφοριών ανάλογα με το αν είναι έρευνα ή αν είναι απλώς αποθήκευση στοιχείων, συγκέντρωση στοιχείων ώστε να είναι αυτά διαθέσιμα για κάποια περίοδο, για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δεν πιστεύω και δεν θέλω τώρα να αφήσω καμιά παρεξήγηση, δεν πιστεύω πως είναι δυνατόν να μειωθεί ο σωρός του άχυρου το μηδέν, ώστε να μένει μόνη η βελόνα. Αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και μας μας απασχολεί αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον όγκο των στοιχείων, των άσχετων στοιχείων, των αθώων στοιχείων, στο μήνυμα ώστε να μπορεί ο κόσμος να είναι ήσυχος ότι μαζί με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές δικλείδες τα δεδομένα τους δεν θα εκμεταλλευτεί κανείς για άλλους σκοπούς. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό να πούμε είναι πως ο σωρός των άχυρων εκτός από τη βελόνα παραμένει ανώνυμος και κλειστός και δεν γίνεται έρευνα σε αυτόν εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, συγκεκριμένος σκοπός και μια έρευνα για κάποιον άνθρωπο συγκεκριμένο, για κάποιο άτομο ή άτομα. Δεν γίνεται εξόριξη στοιχείων και τώρα πώς λειτουργεί το SWIFT σήμερα. Υπάρχει ένα σερβερ για τα βορειοαμερικανικά στοιχεία, ένας ευρωπαϊκός σερβερ για τα ευρωπαϊκά στοιχεία και το υπόλοιπο του κόσμου επιλέγει που θα βάλει τα στοιχεία του. Οπότε, η λαϊκή δημοκρατία της Ιουρτάνε της, θα, θα αποφασίσει πού θα μπουν τα στοιχεία της. Τώρα, αν υπάρχει έτοιμα από τις ΕΠΑ για συγκεκριμένα στοιχεία, εδώ βρίσκονται και εκεί, είναι και που προκύπτει το πρόβλημα. Εσείς ζητήσατε ειδικά μια υποχρέωση για παροχή, μάλλον αναζήτηση προηγούμενης έγκρισης από την Ένωση πριν την μεταφορά στοιχείων που βασίζονται στα στοιχεία TFTP προς τρίτες χώρες. Αυτό το σημειώνω. Είναι ένα θέμα ειλικρινά όπου πιστεύω πως οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το τα στοιχεία TFTP προστίθενται σε ένα σωρό άλλα στοιχεία και οδηγούν σε ενδιαφέρον για την διερεύνηση ενός ή την έρευνα για ένα συγκεκριμένο άτομο. Και αυτά τα στοιχεία είναι που κανονικά μέσα στις διαδικασίες τις αντιτρομοκρατικές αν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ή ακόμα και οι δυνάμεις αντικατασκοπίας μπορούν να μοιραστούν τέτοιες πληροφορίες. Δηλαδή είπαμε με κάποια ξένη χώρα. Θα, βέβαια τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιέχουν λίγα στοιχεία TFTP. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ποια αναλογία στοιχείων TFTP θα χρησιμοποιηθεί γενικότερα. Άρα λοιπόν με αυτές τις συνθήκες το να ζητηθεί προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για αυτό που οι Αμερικανοί θεωρούν κανονική φυσιολογική διεθνή συνεργασία στην τρομοκρατική τους εργασία το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εντάξει το άκουσα, θα το συζητήσουμε και θα σας πούμε τι θα συμβεί ε, σε αυτό το χρόνο. Για την κυρία Τζίπελ, να πω ότι κατάλαβα ότι θα πρέπει να μεταφέρω τόσο γίνεται πιο λίγα στοιχεία. Αυτή είναι και η δική μας πρόθεση. Και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να σας ικανοποιήσουμε τελικά να σας πω σε εσάς που στην κυρία Ιντεβελ που κάθεστε δίπλα, κάθεστε δίπλα μας πως υπάρχει κάτι που τα διέπει όλα αυτά. Είναι μια ιδέα ότι, που, που, που, ελπίζω θα είναι σαφής για τους αναγνώστες της σχεδίου εντολής, ότι δηλαδή θα, αναφέρει, θα αναφέρεται σε ολόκληρο το κείμενο, είναι ένας ε, νόμος και βεβαίως είναι και το βασικότερο κομμάτι της επιχείρησης την οποία εμείς θα κάνουμε. Οπότε ναι και πάλι δεν θα σας αναφέρουμε οτιδήποτε δυσανάλογο. Στον κύριο Μπουζουτήλ. Να πω ότι ναι, έχουμε μάθει τα μαθήματά μας. Φυσικά και τα προβλήματα κρύβονται στις λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες ε, θα προκύψουν με τις διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, αλλά δεν έχει κανείς νομίζω από την πλευρά μας αμφιβολία για το είδος των θεμάτων που σας ανασυχούν και που θέλατε να δείτε στην τελική συμφωνία. Εσείς θέλετε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για την ε, αποκατάσταση. Είπατε ότι ο χρόνος είναι σημαντικός αλλά όχι και ε, απόλυτος. Η αποκατάσταση είναι ένα άλλο θέμα, δηλαδή ξεκινάμε από τα ε, σαφή προϋπόθεση πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους Αμερικανούς, σας τις είπα. Και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων, των Ευρωπαίων πολιτών είναι η προστασία των δεδομένων ένα θεμελιώδες δικαίωμα, δεν είναι διαπραγματεύσιμο, δεν μπορούμε να το διαπραγματιστούμε ούτε και να το ε, παζαρέψουμε σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Άρα λοιπόν θα επιμείνουμε ότι η θεμελιώδης αρχή, ότι δηλαδή έχουν όλο το δικαίωμα να πάνε σε ένα δικαστήριο και να διαμαρτυρηθούν κατά κάποιας διοίκησης, διοικητικής αρχής ε, και τα λοιπά θα πρέπει να ισχύει. Ξέρουμε το νόμο περί ιδιωτικής ζωής που είναι ε, που περιέχει στοιχεία διακρίσεων και φυσικά οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε δίκαια. Τώρα, αν θα έχουμε αποτελέσματα μέχρι το καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα αλλάξει καμιά νομοθεσία, αλλά σίγουρα θα περιμένουμε οι Αμερικανοί ομολογοί μας να δείξουν κατανόηση για το θέμα και να δώσουν με όποιο τρόπο γίνεται το δικαίωμα αμφισβήτησης στο δικαστήριο με τον φυσιολογικό τρόπο όπως θα περίμενε κανείς από οποιοδήποτε δημοκρατικό σύστημα την χρήση την κατάχρηση των στοιχείων που έχουν δοθεί από πλευράς τους. Συγγνώμη που μακρηγόρησα κάπως, ελπίζω να απάντησα στις κύριες ερωτήσεις. Είναι μια νέα αρχή μια νέα συνθήκη, ένα νέο πολιτικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Κανένας δεν έχει αμφιβολία περί αυτού. Ελπίζουμε πως η εντολή θα υιοθετηθεί και θα μας δώσει σαφή κατεύθυνση, σαφείς οδηγίες. Θα λαμβάνουμε υπόψη την παράλληλη πολιτική εντολή που προκύπτει από αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρουμε πως στο τέλος θα πρέπει να σας δώσουμε κάτι το οποίο θα δεχτείτε. Και θα διαπραγματευτούμε καλή την πίστη από αυτές τις βάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φόλ για όλες τις πληροφορίες και την προθυμία που δείξατε στις διαπραγματεύσεις για τις επερχόμενες ε, διαπραγματεύσεις. Κύριε Άντμπραχτ, ε, μια ερώτηση σύντομη από εμάς. Μήπως η νομική υπηρεσία θα μπορούσε να εξετάσει κατά πόσον εμείς μπορούμε ως Κοινοβούλιο να ζητήσουμε την γνωμοδότηση του ΔΕΚ για την εντολή και τη σχέση της εντολής ε, με τη συνθήκη πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να περιμένουμε μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων για να υπάρχει μία άποψη του ΔΕΚ για το πλαίσιο και για το αν ε, το, συνταγμα, συνταγματικό πλαίσιο είναι θεμητό ή όχι. Υπάρχει κάποια τέτοια δυνατότητα γιατί στο τέλος θα και θα πρέπει να αποφασίσουμε γρήγορα. Και νομίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας επιβάλλει την υποχρέωση προστασίας του συνταγματικού μας πλαισίου. Το σημειώνουμε αυτό το διαδικαστικό αίτημα του κυρίου Άλμπερτ η συνθήκη όντως περιλαμβάνει μια τέτοια νομική δυνατότητα. Το άρθρο 218 παράγραφο 11 Η νομική υπηρεσία, ο κ. Περίλο θέλει να το σχολιάσει. Πρόεδρε, όπως είπατε, η συνθήκη όντως περιλαμβάνει μια διάταξη, το άρθρο 18, 2.18 συγγνώμη παραγραφό 11 που επιτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από το ΔΕΚ να γνωμοδοτήσει επί των λεγόμενων προβλεπόμενων συμφωνιών. Η νομολογία του ΔΕΚ περιέχει περιγραφή τι είναι προβλεπόμενες ε, συμφωνίες. Κατά την άποψή μου δεν νομίζω να υπάρξει δυσκολία στο να λάβουμε υπόψη το ενδεχόμενο να ακούσουμε τη γνωμοδότηση του ΔΕΚ για την συμμόρφωση της προβλεπόμενης αυτής συμφωνίας με τη συνθήκη. Αυτό βέβαια είναι ένα πολιτικό ζήτημα Η νομική βάση πάντως αυτή της δυνατότητας υπάρχει στη συνθήκη και την άποψη αυτή μπορεί να τη ζητήσουν τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Θα το εξετάσουμε, το σημειώνουμε τέλο πάντων. Αυτά προς το παρόν. Κλείνουμε την πρωινή συνεδρίαση. καλύψαμε την προβλεπόμενη μερίσια διάταξη αυτή της πρωινή συνάντηση, Προτείνω να μείνουν εδώ οι συντονιστέ για να γίνει συνάντηση συντονιστών και κλεισμένων των θυρών παρόντος καταρχήν του Γενικού Διευθυντού κ. Φόλ για τον διατραντικό διάλογο και η υπόλοιπη μερίσια διάταξη θα είναι και κλεισμένο των θυρών απόλυτα. Θα ξεκινήσουμε ξανά στις 4.30 το απόγευμα μετά την ε, ολομέλεια του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου για την ε, Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συνοβουλίου. Διακόπτουμε λοιπόν μέχρι τις 4.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ.